Καλημέρα σας ε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ε, η ακρόαση για το κοσυφοπαίδιο θα γίνει αύριο το πρωί στις 9 και η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 11.45. Ε, έχουμε και κάποιες άλλες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Θα έχουμε τη συζήτηση για το μέσο της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει μια συζήτηση για τους υπόλοιπους μηχανισμούς και στις 5 θα γίνει μια συζήτηση για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες Αν συμφωνείτε λοιπόν με τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και περνάμε και στην έγκριση των πρακτικών. Διάβασε κανείς τα πρακτικά, υπάρχουν ενστάσεις, αλλιώς ε, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Εγώ δεν έχω τίποτα να ανακοινώσω περαιτέρω. Για να περάσουμε λοιπόν απευθεία τώρα στην ανταλλαγή απόψεων με τον ε, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, ε, τον ε, κύριο Ραντάμε Λαμάμρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι αυτές οι ανταλλαγές απόψεων ε, για την ειρήνη και την ασφάλεια της Αφρικανικής Ένωσης είναι σημαντικές. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε εντατικές ανταλλαγές απόψεων, ιδίω ε, λόγω των ε, ε, σειράξεων στο Σουδάν και στις δύο πλευρές, στο Μαλί, τη Γουινέα Μπισάου. Κύριε Πρέσβη, γνωρίζω ότι σας περιμένει πάρα πολύ και σκληρή δουλειά και φαντάζομαι ότι θα έχετε αρκετά πράγματα να κάνετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αφρικανικής Ένωσης ε, προκειμένου να προλάβει τις σειράξεις ε, και να βρεθούν ε, ειρηνικές λύσεις. Ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ο ρόλος του συμβουλευτικού πάνελ και οι οργανώσεις της Περιφερειακής Συνεργασίας της Αφρικανικής Ένωσης και θα θέλαμε να ξέρουμε πώς μπορεί η, Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει και αυτή την υποστήριξή της για την επίλυση των προβλημάτων στην ε, Αφρική. Σας δίνω λοιπόν το λόγο και ελπίζω να έχουμε μια καρποφόρα συζήτηση. Σας ευχαριστώ εγώ, ε, εσάς και τα μέλη της Επιτροπής σας που με προσκάλεσατε. Με χαρά ξανάρχομαι ε, Στο παρελθόν έχω ανταλλάξει, ανταλλάξει απόψεις με την Επιτροπή και με την Υποεπιτροπή σας και διατηρώ άριστες αναμνήσεις. Αυτές οι επαφές αποτελούν και ενθάρρυνση να συνεισφέρω ακόμα περισσότερο σε αυτό τον διάλογο στο πλαίσιο της ε, προνομιακής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αφρικανική Ένωση. Όπως γνωρίζετε, η στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στις δύο ε, οικοδομείται και έχει ήδη να επιδείξει και καρπούς. Τα, οι κοινέ συνοδοι Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρικανική Ένωση από το Κάιρο, τη Λισαβόνα και τελευταία στην Τρίπολη έχουν πάρει συγκεκριμένε αποφάσεις για την οικοδόμηση αυτής της σχέσης. Βρισκόμαστε στην πέμπτη συμβουλευτική συνεδρίαση ε, του Συμβουλίου Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης με την Πολιτική Επιτροπή και, Πολιτική και ε, ε, Επιτροπή Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερη γιατί εμείς γιορτάζουμε τα 10 χρόνια της δημιουργίας μας. Η, αφρικανική, κοινή αφρικανική δράση βέβαια ξεκίνησε το 1963 στο πλαίσιο της οργάνωσης της Αφρικανικής Ενότητας, όμως ε, πριν από 10 χρόνια θεωρήσαμε πως ε, ήρθε η ώρα η κοινή αφρικανική δράση να αποκτήσει νέες προοπτικές, νέες φιλοδοξίες και αυτό μέσω καινούριων κειμένων, ε, εργαλείων και δομών. Η Αφρικανική Ένωση λοιπόν παρέλαβε την σκητάλη από την, ε, ε, την έννοια αφρικανική δράση και βέβαια ε, κληρονόμησε και τις αδυναμίες της. Η, παρ' όλα αυτά είναι μια ε, καινούργια οργάνωση και ποιοτικά ε, έχει ευρύτερο πεδίο δράσης. Η, το στρατηγικό όραμα της Αφρικανικής ε, Ένωσης προβλέπει τέσσερις πυλώνες. Πρώτον, ειρήνη και ασφάλεια ως ανάγκη, ως υποχρέωση, υποχρεωτική προ, ε, προϋπόθεση για τους υπόλοιπους τρεις πυλώνες, δεύτερος πυλώνας, κάτι που μας ξεχωρίζει από άλλες οργανώσεις, οι κοινέ αξίες, δημοκρατία, καλή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που δεν υπήρχε στην ενή αφρικανική δράση, στους ε, κανόνες δράσης της. Τρίτον, συνεργασία και ολοκλήρωση της Υπήρου. Και τέταρτος πυλώνας ε, θεσμικές και ανθρώπινες δυνατότητες και θεσμοί ε, Αφρικανικό Δικαστήριο, Αφρικανικό Κοινοβούλιο και άλλοι θεσμοί που δημιουργήθηκαν για να προωθήσουν την ολοκλήρωση στην Αφρικανική Ήπειρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια και την ειρήνη, της, τον οποίο έχω αναλάβει εδώ και τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο της πρώτης ε, εκλεγμένης θητείας, ε, θητείας κατόπιν εκλογών ε, η, το, η γκάμα των δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνει την πρόληψη ε, διαρθρωτική καταρχήν των συγκρούσεων δηλαδή την αντιμετώπιση των λόγων που δημιουργούν τις συγκρούσεις των αιτίων δηλαδή μετά έχουμε την ε, ε, εμβάθυνση της ε, ειρήνης από τη στιγμή που εφαρμόζονται προγράμματα ειρήνευσης και λαμβάνονται μέτρα για κάθε μία από τις περιπτώσεις συγκρούσεων ενδεχομένω. Μετά έχουμε μία διαφορά σε σχέση με την οργάνωση των Αφρικανικών κρατών. Ε, η οργάνωση των Αφρικανικών κρατών ε, βασίζεται στην αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις. Η Αφρικανική Ένωση όμως είναι η πρώτη διεθνής οργάνωση, ο πρώτος διεθνής οργανισμός που ε, στα βασικά της κείμενα έχει καταγράψει την ευθύνη προστασίας. Ε, η συντακτική πράξη της Αφρικανικής Ένωσης ε, βασίζεται στην μία πάθεια. Οπότε προβλέπει την παρέμβαση ε, της Αφρικανικής Ένωσης σε περίπτωση συγκρούσεων έστω και στρατιωτική παρέμβαση στην περίπτωση που η ΑΒ χώρα, στην ΑΒ χώρα παρατηρείται, παρατηρούνται σημαντικές και βαριές ε, ε, παραβιάσεις συγγνώμη, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ των βασικών αρχών της Αφρικανικής Ένωσης που κληρονομήσαμε από την ε, προηγούμενη μας οργάνωση είναι ε, το απαραβίαστο των συνόρων. Αυτή η αρχή έχει συμπεριληφθεί στη συντακτική πράξη της Αφρικανικής Ένωσης δεν αποτελεί πλέον όπως παλιά ένα ψήφισμα. Ε, η συντακτική συνθήκη ε, της Αφρικανικής Ένωσης την προβλέπει αυτήν αρχή. Αρχή η οποία εμπνέει και όλες τις ε, προσπάθειες ολοκλήρωσης της Αφρικανικής Υπήρου αντίθετα με τάσεις κατακαιρματισμού που μπορεί να υπάρχουν. ε, για παράδειγμα η θερμή πραγματικότητα του Βόρειου Μαλή. Μεταξύ των άλλων καινοτομιών είναι επίσης ότι ε, δεδομένου ότι όλες οι καινούριες κρίσεις και καινούριες συγκρούσεις στην Αφρική έχουν άμεσα ή έμεσα σχέση με την διακυβέρνηση έχουμε ε, εξετάσει και εξετάζουμε πολύ προσεκτικά όλα τα θέματα διακυβέρνησης και δεν έχουμε μόνο βασικές γενικές αρχές αλλά και θεσμούς και όργανα έτσι ώστε να προωθήσουμε την καλή πολιτική, οικονομική ε, και επιχειρηματική διακυβέρνηση ε, για παράδειγμα αγώνας εναντίον της διαφθοράς. Η εργαλειοθήκη που διαθέτουμε ε, είναι όλο και πιο πλούσια Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αφρικανική αρχιτεκτονική ε, και ασφάλειας. Πρόκειται για ένα συνολικό σύστημα συλλογικής ασφάλειας που έχει ως στόχο όχι μόνο την πρόληψη των συγκρούσεων αλλά και την επίλυση των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των αιτίων τους έτσι ώστε να μην ξαναεμφανιστούν στο μέλλον. Ε, σε ό,τι αφορά τι συγκρούσει και τι κρίσει σχετικέ με την διακυβέρνηση, έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία αυτών των συγκρουσιακών καταστάσεων ε, ε, έχει σχέση με την ε, εξισορρόπηση ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, ανάμεσα στις ελευθερίες και, και την πραγματικότητα. Ε, υπάρχουν ανισορροπίες, ε, υπάρχουν ε, δυσκολίες οι οποίες έγκυται στην απουσία αναλογικότητας ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Το κέντρο συνήθως έχει μεγαλύτερη ισχύ από την περιφέρεια και από την άλλη μεριά έχουμε την ενότητα και τις διαφορές και τη διαφορετικότητα, δηλαδή η ενότητα πολλές φορές γίνεται εις βάρος της διαφορετικότητας. Και αυτό δημιουργεί ε, διασπαστικές τάσεις ή παρεμβατικές τάσεις. Θα έχετε παρατηρήσει σίγουρα ότι στην σημερινή Αφρική σχεδόν όλες οι κρίσεις και οι συγκρούσεις είναι εσωτερικές. Στην πραγματικότητα σχεδόν δεν έχουμε πλέον συγκρούσεις ανάμεσα σε γειτονικέ χώρες. Δεν έχουμε ε, δηλαδή πολέμους και συγκρούσεις ε, για αλλαγή των συνόρων ή για απόκτηση ε, πόρων από γειτονικέ χώρες. Οι συγκρούσεις πλέον περιορίζονται στο εσωτερικό κάθε χώρας. Όμως βέβαια πολλές φορές παίρνουν αυτές οι συγκρούσεις ε, περιφερειακές ε, διαστάσεις είτε εξαιτία παρεμβάσεων από το εξωτερικό είτε εξαιτία παραγόντων που συνδέονται με εθνοτικές ομάδες που ξεπερνούν τα σύνορα. Να σας ενημερώσω εν συντομία για τις ε, καταστάσεις ε, συγκρούσεων που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Καταρχήν είναι ένα θετικό σχόλιο που πολλές φορές αγνοούμε. Σήμερα έχουμε πολύ λιγότερες συγκρούσεις και πολύ λιγότερα θύματα από ότι στην τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. Θυμάστε ποια ήταν η κατάσταση στις μεγάλες λίμνες Θυμάστε ποιες ήταν οι καταστροφικές συνέπειες του, της γενοκτονίας της Ρουάντα. Δέκα χρόνια μετά έχουμε λιγότερες συγκρούσεις, λιγότερα θύματα στην Αφρική. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας χαροποιεί, παρόλο ότι και πάλι έχουμε υπερβολικά πολλές συγκρούσεις και υπερβολικά πολλά θύματα. Ε, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσουμε ε, ανθρώπινες ζωές, ε, πρέπει να το κάνουμε Στόχος είναι η Αφρική σε ειρήνη με τον εαυτό της και με τους άλλους. Αυτό είναι και το σύνθημά μας. Τα εγκάρσια ζητήματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην Αφρική ε, περιλαμβάνουν την ε, θαλάσσια πειρατεία, την τρομοκρατία, ε, όλο και περισσότερες ομάδες ε, που έχουν ως στόχο τη διάσπαση των χωρών τους ε, και παρατηρήστε ότι από τον, κόλπο του Άντεν στη Σομαλία μέχρι τον κόλπο της ε, Γουινέας στην δυτική ακτή της Αφρικής έχετε ένα τόξο κρίσεων που θα μπορούσαν να περιγραφούν ως λεωφόρος των συγκρούσεων. Ε, είναι ένα τόξο Δύση Ανατολή, στην κατεύθυνση Δύση Ανατολή, που αποτελεί πραγματικό πρόβλημα ε, και εμπόδιο στην ε, πρόθεση της συνολικής ασφάλειας στην Ήπειρο. Να προσθέσω ότι το διασυνοριακό έγκλημα έχει μια έκφανση ιδιαίτερα σοβαρή πέραν της πειρατείας και της τρομοκρατίας που είναι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Αναμφίβολα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ουσιών στην Αφρική δεν είναι πλέον ε, μόνο ένας ε, κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών, που ισχύει βέβαια, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, αφισβητεί ταυτόχρονα ε, και υποσκάπτει την λειτουργία της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών. Οπότε αποτελεί όλο και περισσότερο κίνδυνο για την περιφερειακή ασφάλεια όλη η Αφρική, ε, η Δυτική Αφρική, ε, αποτελεί θύμα αυτής, αυτού του λαθρεμπορίου. Ε, η Δυτική Αφρική αποτελεί κυρίως ε, ένα σημείο διαμετακόμισης τράζη των ναρκωτικών παρόλο που ένα τμήμα των ναρκωτικών μένουν, μένει εκεί και επηρεάζει τη ζωή ιδιαίτερα των νέων ή το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών αυτή τη στιγμή πλέον πρέπει να θεωρείται ως απειλή για την ασφάλεια και την ε, ειρήνη στην περιοχή της Αφρικής. Η... Τελικά η απειλή είναι μήπως και στη Δυτική Αφρική δημιουργηθούν ναρκοκράτη ε, όπου τα δίκτυα θα έχουν πλέον την εξουσία, δίκτυα που ξεκινούν από την Νότια Αμερική και προσπαθούν ε, να διασφαλίσουν τη θέση τους ε, μεταξύ Νότιας ε, Αμερικής και Ευρώπης που αποτελεί την, την αγορά τους. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πρόβλημα. Τώρα σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες καταστάσεις δεν θα τις περιγράψω με λεπτομέρεια αν μου επιτρέπετε αργότερα μου θέσετε ερωτήματα μπορώ να δώσω περισσότερα στοιχεία. Έχουμε, ε, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη η περιοχή των μεγάλων λιμνών. Ε, για παράδειγμα, ε, στα ανατολικά της Δημοκρατίας του Κονγκό, όμως και στο Μπουρούντι, παρόλο ότι ε, τα πιο θερμά μέτωπα είναι σε άλλα σημεία της Επίρου Πρέπει να ε, μην αγνοήσουμε την κατάσταση στην, ε, στις Μεγάλες γιατί μπορεί να χειροτερεύσει. Ιδιαίτερα δυσχερής είναι η κατάσταση επίσης και μπορεί να καταλήξουμε και σε τραγωδία αν δεν προσέξουμε, είναι η κατάσταση στο μεταξύ Σουδάν και Νότιου Σουδάν. Ε, στην Αντίσα Μπέβα ξεκίνησαν ξανά οι διαπραγματεύσει υπό την αιγίδα του πάνελ υψηλού επίπεδου της Αφρικανικής Ένωσης με πρόεδρο το κύριο Μπέκι, πρώην πρόεδρο της ε, Νότιας Αφρικής. Ε, το κέρα της Ανατολικής Αφρικής είναι επίσης πολύ ευαίσθητο. Έχουμε καλές εξελίξεις στη Σομαλία υπέρ της δράσης της διεθνούς κοινότητας με, με την υποστήριξη τη συνεχή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρικανική Ένωση ε, με χρηματοδότηση και ξαναστήσιμο ε, του, της ε, Σομαλίας. Ε, στις 20 Αυγούστου θα τελειώσει μάλλον η μετάβαση σε ένα πιο δημοκρατικό καθεστώς με σύνταγμα και αυτό μας ε, δημιουργεί ελπίδες. Ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα αποτελέσει παράδειγμα για την δράση της διεθνούς ε, κοινότητας και στο μέλλον. Για την επίλυση προβλημάτων τα οποία φαίνονται ανεπίλητα. Μετά, στο Σάχελ το Σάχελ είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ε, παλιότερα είχαμε τα αποστήματα των μεγάλων λιμνών και του κέρατος της ε, Ανατολικής Αφρικής. Πλέον το Σάχελ παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ των συγκρούσεων ε, διότι εξαιτίας μάλλον της, ε, των προβλημάτων διακυβέρνησης, ε, των ανθρωπιστικών προβλημάτων, περιβαλλοντικών προβλημάτων, τρομοκρατίας, ναρκωτικών κλπ. Υπάρχει μια ένα ολόκληρο σκηνικό, ένα κοκτέιλ δυσκολιών σε όλη αυτή την περιοχή δυσκολίες οι οποίες ξεπερνούν την δημοκρατία του Μαλή και αποτελούν πλέον περιφερειακό πρόβλημα που μάλιστα ξεπερνάει και τη Δυτική Αφρική γιατί εμπλέκει και ε, και άλλες χώρες, ε, εμπλέκει άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής ή της Κεντρικής Αφρικής. Υπάρχει μια κατηγορία συγκρούσεων τις οποίες μπορούμε να θεωρήσουμε παγωμένες διότι δεν έχουν ε, εξωτερικές εκδηλώσεις βίας ούτε όμως ε, και σημαντική πρόοδο προς την επίλυσή τους. Για παράδειγμα, Αιθιοπία-Ερυθρέα, Τζιμπουτή-Ερυθρέα, καθώς επίσης και η διαδικασία διαδικασία της ολοκλήρωσης ε, της ε, από ε, απεικιοποίηση της Δυτικής Αφρικής με τις ε, ε, της Δυτικής με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με την διοργάνωση του δημοψηφίσματος που έχει προβλεφθεί. Εκεί σε αυτές τις τρεις περιοχές έχουμε πραγματικά διέξοδο. Ε, για την πρόθεση της ασφάλειας και της ειρήνης έχουμε και ένα καινούριο εργαλείο, ε, την ενισχυμένη ε, πρωτοβουλία συνεργασίας με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του, των Ηνωμένων Εθνών. οι αφρικανικές χώρες αποδεικνύουν με αυτόν τον τρόπο ότι ε, παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα κάθε φορά ε, μέτρα ε, σε αφρικανικό επίπεδο ή σε πιο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κάθε φορά στην επίλυση των διαφορών. Εν συντομία να σας πω, να σας μιλήσω για την θετική και επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό που ονομάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως Αφρικανική Άνοιξη. Ε, εμείς μιλούμε για λαϊκή εξέγερση ή για επανάσταση πιο πολύ. Είναι μια δυσχερής διαδικασία δημιουργίας δημοκρατικών θεσμών μέσω εκλογικών αναμετρήσεων. Για την Αφρική αυτό είναι κάτι πολύ καινούριο, δίνει πολλές ελπίδες για παράδειγμα στη Λιβύη που ετοιμάζει τη συντακτική της συνέλευση. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία ε, μετασχηματισμού στη Βόρεια Αφρική, η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή και ε, εμείς έχουμε καθήκον να παρακολουθήσουμε από κοντά την κατάσταση, να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες και να αποφύγουμε ε, την, τον εκτροχιασμό της. Δεν εργαζόμαστε μόνοι μας, εργαζόμαστε με εταίρους πιστούς, στρατηγικούς εταίρους. Για παράδειγμα με την, με την Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησα για αυτή τη ε, σχέση. Νομίζω ότι είναι μια σχέση όριμη πλέον. Ε, με ουσία σημαντική για να λειτουργήσει η αρχιτεκτονική ασφαλείας και ειρήνη στην Αφρικανική Ήπειρο και χαιρόμαστε για αυτή τη συνεργασία και την συνεχή υποστήριξη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή η συνεργασία έχει φτάσει σε ένα πολύ αξιόλογο επίπεδο. Να πω μόνο ότι τους πρώτους μήνες του 2012 ε, το ψήφισμα 2036 του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Σομαλία ε, μέσω του που δέχεται την στρατηγική πολιτική, τη στρατηγική της Αφρικανικής Ένωσης ε, για την ε, ενίσχυση της ε, ασφάλειας στην Σομαλία ή το 2046 της Δευτέρας Μαΐου για το Σουδάν και, Σουδάν και το Νότιο Σουδάν που ψήφισμα το οποίο επαναλαμβάνει λέξη προς λέξη ε, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης είναι αποδείξη αυτής της ε, οριμότητας της συνεργασίας. Ε, η πεντηκοστή επέτειος από την δημιουργία της οργάνωσης της Αφρικανικής Ένωσης θα διορταστεί του χρόνου με την πεντηκονταετία από την ανεξαρτησία ορισμένων χωρών της Υπήρου μας. Ο Παναφρικανισμός παραμένει πολύ ζωντανός ε, στο μυαλό και στην πολιτική των Αφρικανών με στόχο την αναγέννηση της Αφρικανικής Υπήρου ε, οικοδόμηση πάνω στα κεκτημένα ε, διόρθωση των αδυναμιών και ελπίζουμε ότι η Αφρική θα προχωρήσει, θα προοδεύσει εξασφαλίζοντας ε, ε, πλήρως την εφαρμογή των αρχών που συμμερίζεται με την, με την διεθνή κοινότητα, αρχών που ε, θα μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε το δρόμο της ανάπτυξης, της πρόοδου προς μια Αφρική ειρηνική υπεύθυνη στη διεθνή κοινότητα και ευημερούς. Ευχαριστώ. Ich bedanke mich sehr σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ από την πλευρά μου. Για αυτή την παρουσίαση η οποία θα αποτελήσει ε, τροφή προς συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, παρουσίασή σας. Όπως είπατε, η Αφρικανική Ένωση είναι πολύ σημαντικός εταίρος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως όπως μας υπενθυμίσατε, υπάρχουν κάποια πολύ ανησυχητικά στοιχεία. Εγώ θα θέλω να αφαιρθώ σε δύο από αυτά τα κρίσιμα της κρίσης, αν θέλετε. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του Σουδάν και του Νοτίου Σουδάν. Βεβαίως χαιρόμαστε που ξεκίνησαν ξανά οι διαπραγματεύσει. Ε, πριν από μία εβδομάδα, ωστόσο, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, είπαμε ότι μας προβληματίζει ιδιαίτερα η επανέναρξη των ε, βομβαρδισμών την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, βεβαίως, είδαμε ότι η Αφρικανική Ένωση δεν ε, καταδίκασε τους βομβαρδισμούς που αυτό είναι ένα μέσο για να ε, ενθαρρύνεται το, το Νότιο Σουδάν να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις ή νομίζετε ότι από εδώ και πέρα αυτό θα είναι ε, ένα εργαλείο που μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή τρεις μέρες βομβαρδισμού και μετά επανερχόμαστε στις ε, διαπραγματεύσεις. Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο σκοπός αυτών των βομβαρδισμών από τον Νότιο Σουδάν. Δεύτερη παρατήρηση για τη Σομαλία. Την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ και συνάδελφοί μου είδαμε ότι ε, ε, οι Αφρικανικές Ένωσες έχουν πολύ σημαντικές ε, δυνάμεις ό,τι αφορά την Αυγόε που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα στην Σομαλία ε, για την δημιουργία ενός ε, ανθρωπιστικού διαδρόμου μέχρι το Μογκαντήσου. Βεβαίω και πρέπει να συγχαρούμε τις στρατιωτικές δυνάμει για την επιτυχία του. Το ερώτημά μου, θεωρείτε ότι αυτός ο διάδρομος ε, θα διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα. Θα μπορούσε να είναι μια να είναι μια ενέργεια που θα κρατήσει. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Γκόμες, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη, κύριε Επίτροπε, για τη διεξοδικότητα παρουσίασή σας. Πολύ εύστοχα τα στοιχεία που μας είπατε και εγώ προσυπογράφω τις ερωτήσεις που έθεσε ο συνάδελφος, αλλά θα ήθελα να μας εξηγήσετε και τη στάση της Αφρικανικής Ένωσης για την κατάσταση στο Μαλί και στη Γουινέα Μπισάου. Διότι οι βασικές αρχές που μας περιγράψατε, οι οποίες είναι βεβαίως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση, αλλά και οι προκλήσεις ε, στις οποίες σταθήκατε, για το γεγονός ότι κάποια κράτη είναι αδύνατο να κυβερνηθούν. Και τελικώς ε, είναι ε, έρμεο σε όλες τις μορφές το οργανωμένο έγκλημα, κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών και όλα αυτά αμφισβητούνται και από την δράση του ΕΚΟΑΣ. Ο ΕΚΟΑΣ υποτίθεται ότι είναι μια περιφερειακή οργάνωση στη Δυτική Αφρική, ε, που υπόκειται βεβαίως στην Αφρικανική Ένωση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δρά αυτή τη στιγμή ο ΕΚΟΑΣ, ο οποίος ουσιαστικά δημιουργεί απικίε και υποστηρίζει ε, όλα αυτά τα κινήματα ε, που γίνονται για την ανατροπή κυβερνήσεων, ουσιαστικά έρχεται σε αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει η Αφρικανική Ένωση αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη και όσα θα έπρεπε να πρεσβεύει. Και νομίζω ότι στην περίπτωση της Γουινέα Μπισάου είναι σίγουρα σε αντίθεση με το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση να συνεργάζονται περισσότερο, έχοντας πάντα και κατά νου αυτούς τους διαδρόμους ε, οργανωμένου εγκλήματο, τους οποίους μας ε, παρουσιάσατε και που φαίνεται ότι πλέον εκτείνονται από Ανατολάς προς Δυσμάς ε, σε όλη την Αφρική. και είπατε ότι ε, φαίνεται ότι αυτό το οργανωμένο έγκλημα ε, αποτελεί πληγή για τους ε, λαούς της Αφρικής. Θα ήθελα επίσης να μας ε, πείτε λίγα περισσότερα πράγματα και για το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Ξέρω ότι μας είπατε ότι η Αφρικανική Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα ψηφίσματα της ε, ε, των Ηνωμένων Εθνών ε, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, που είναι σίγουρα η περίπτωση της Δυτικής Σαχάρας, ΕΛΟ. Εδώ όμω βρισκόμαστε ενώπια μια κατάσταση όπου ε, σαφώ το διεθνέ δίκαιο. Και όπω είπατε κι εσεί, ο επίτροπο Κρίστοφερ Ρο, πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δεν έγινε δεκτός από το Μαρόκο. Αποτελεσματική Αφρικανική Ένωση στο θέμα αυτό. Να σας πω βεβαίω ότι θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη για την αδράνεια αυτή την οποία εμφανίζει το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά το θέμα είναι ότι πρόκειται για αφρικανικό πρόβλημα και θα πρέπει ε, τα ηνία σε αυτό το θέμα να το έχει η Αφρικανική Ένωση. Και δεν βλέπω να ε, δραστηριοποιήσετε. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε λοιπόν και αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω ότι Παρεμπιπτόντω, είχαμε συναντηθεί και στη Βιέννη και χαίρομαι ιδιαίτερα που σα ε, ξαναβλέπω. Θεωρώ ότι η διεξοδικότατη παρουσίασή σα ακριβώς επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι για μας ε, να ανταλλάσσουμε απόψεις ε, πιο τακτικά, σε περισσότερο πολιτικό επίπεδο και να εμβαθύνουμε και περισσότερο. Και νομίζω ότι μας έχετε δώσει τροφή για σκέψη σήμερα μετά όσα μας είπατε. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω καταρχάς για τη Δυτική Σαχάρα. Εχθές το απόγευμα είχαμε μία εκδήλωση ε, με πάρα πολύ κόσμο, δεν υπήρχε θέση ελεύθερη. Είχαμε και 50 ορθίους και το θέμα προς συζήτηση ήταν η Δυτική Σαχάρα. Ε, προβλήθηκε και μία ταινία για τη Δυτική Σαχάρα. Αλλά το πιο σημαντικό ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι Ποιο είναι ο πλέον αρμόδιος για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και να ξεκινήσει μια διαδικασία επίλυση του ζητήματος. Εχθές είδαμε εικόνες για το πώς ξεκίνησε το πρόβλημα και είδαμε ότι όλα ξεκίνησαν από μια βάρβαρη εισβολή. ήταν ουσιαστικά μια επινόηση αυτή η σύγκραξη, διότι τέθηκε θέμα κυριαρχίας των ανθρώπων που ζούσαν στην ε, γη τους και επιστροφής της κυριαρχίας. Και θεωρώ ότι όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά των κρατών μελών τους που ορισμένες φορές αποτελούν πρόσκομα για την λογική λύση ενός προβλήματος εντός των Ηνωμένων Εθνών και εκτός, αντιστοίχως το ίδιο αναμένουμε και από εσά, από το δικό σας τον οργανισμό, να λάβει σαφή και θέση και ξεκάθαρη θέση για το θέμα αυτό, διότι αυτό αποτελεί απόδειξη ότι θα πρέπει να επιληθούν τα θέματα στην ε, ε, Αφρικανική Ήπειρο ε, εν γέννη. μπορεί να περιμένουμε να οριμάσει η δημοκρατία στο Μαρόκο, ε, αλλά μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι, ε, και να συνειδητοποιήσουν ακριβώς ότι δεν μπορούν να έχουν μια απικία στην ευρύτερη τους γειτονία ή θα πρέπει να συμβεί κάτι άλλο, το οποίο θα ε, καταδείξει ότι το Μαρόκο είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί επί του ζητήματος και ο συμβιβασμός σημαίνει να ακολουθήσει το νόμο να αποσυρθεί και να δώσει το δικαίωμα στο λαό της Δυτικής Σαχάρας να αποφασίσει μόνος του για το μέλλον του. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι πιο σύντομο και αφορά το θέμα του Νταρφούρ. Το Νταρφούρ επισκιάζεται από τη ε, σύγκρουση μεταξύ ε, Νοτίου και Βορείου Σουδάν. Αλλά δεν ε, ε, πάβει να υφίσταται. Οι διαπραγματεύσεις στην Τόχα δεν οδήγησαν ε, σε επίλυση του προβλήματος για τον Ταρφούρ και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα επανέλθει στο προσκήνιο και θα αρχίσει να μας ε, ενδιαφέρει και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν και κάποια σχόλια από πλευρά σας για τον Ταρφούρ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φανίλσεν. Κύριε Φανίλσεν, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας υποβάλω δύο ερωτήματα. Πρώτον, για το Μαλί. Χθε ε, ο κύριος Φασαβαλάν, πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ε, αναφέρθηκε ε, στην Αφρικανική Ένωση και ζήτησε να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει θέση για την κατάσταση στο Μαλί, το στομότερο δυνατόν. Εξάλλου ήρθε και σε επαφή με τον κύριο Μπονί και με τον κύριο Γουαταρά από τη ΣΥΝΤΕΑΟ. Θα ήθελα να, μου πείτε την άποψή σας για αυτή την ε, σκέψη που εκφράζεται ε, αρκετά συχνά πλέον να υπάρχει μια ε, εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαλί και, και της Αφρικανικής Ένωσης ε, για την ενίσχυση των δυνάμεων της ειρήνης. Ποιος θα ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την άποψη που εκτός από σημαντικό φορέα, ε, εκτός από σημαντικός φορέας ε, σε ανθρωπιστικό επίπεδο έχει τη δυνατότητα να διεξαγάγει ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Τώρα, ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα για την ανθρωπιστική κρίση, την επιστημιστική κρίση. Ε, που στο Βόρειο Μαλί ε, δεν είναι ε, πρόσφατο φαινόμενο γιατί και από το παρελθόν έχουμε περιβαλλοντική κρίση με την ξηρασία και όλα αυτά, αλλά και τώρα αυτό το πράγμα γίνεται, αυτή η κατάσταση χειροτερεύει. Πλέον ε, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και ιδιαίτερα σε ανθρωπιστικό επίπεδο, ιδιαίτερα στον κύκλο του Μποντιαγκαράκ, μια ιδιαίτερα φτωχή ε, περιοχή. Επομένω, από ανθρωπιστική πλευρά ε, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Θα ήθελα επίση να σα ρωτήσω ποιο είναι το αίτημα του MNLA σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ζώνες εγώ εξεπλάγει όταν είδα σε ένα χάρτη το, το, κύκλο του Βόνια που γνωρίζω πολύ καλά Έχω εκπλαγεί λοιπόν, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες ε, σε ό,τι αφορά τα, τα σύνορα που έχουν ε, οριστεί από το απελευθερωτικό κίνημα ε, αυτής της περιοχής. Άλλο ερώτημα πολύ σύντομα. Σας άκουσα να μιλάτε για τις ε, τρέχουσες συγκρούσεις στην Αφρική και είπατε ότι τώρα στην Αφρική είναι, οι συγκρούσεις είναι και διεθνικές. εγώ εκπλήσωμαι από αυτή σας τη δήλωση και δεν συμφωνώ απολύτως. Ε, νομίζω ότι μπορεί ε, να υπάρχουν ε, πρώην αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό βρίσκεται στη βάση της ένοπλης σύραξη στο Κονγκό. Την προηγούμενη εβδομάδα 30.000 ε, άτομα ε, διέφυγαν για να ξεφύγουν από αυτή την ε, ένοπλη σύγκρουση. Δεν μπορούμε λοιπόν, λοιπόν να αρνηθούμε την παρουσία των επιχειρήσεών μας που εκμεταλλεύονται τον φυσικό πλούτο αυτών των χωρών. Ευχαριστώ. Uh, Ο κύριος Τάνοκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ πίσω είμαι. Για το θέμα της Δυτικής Σαχάρας, νομίζω ότι οι δύο συνάδελφοι που σας έφεσαν ερωτήσεις είναι λίγο άδικοι, διότι το Μαρόκο δεν συμμετέχει στην Αφρικανική Ένωση, ακριβώς διότι έχει αναγνωριστεί η Δυτική Σαχάρα από όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην Αφρικανική Ένωση. Είναι ε, η μόνη χώρα που δεν συμμετέχει στην Αφρικανική Ένωση από την Αφρική ακριβώς για αυτό το λόγο. Αναφερθήκατε σε κάποιε παγωμένε σειράξει ε, και τη δημιουργία δύο νέων ε, χαωρών στην Αφρική τα τελευταία χρόνια, ε, το Νότιο Σουδάν. Εγώ ενδιαφέρομαι για το Σομάλιλαν, το οποίο είναι ανεξάρτητο εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχει ο Αλσαμπάμπ, υπάρχει η, η Τζιχάντη, η τρομοκράτες και περιορίζεται η δημοκρατία. Είναι καλές οι ειδήσει από το Σομάλιλαντ και υπάρχουν κάποιες ε, ειδήσει ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή η οποία καταπίεσε την ε, περιοχή. Υπήρχε μία εβδομάδα στην οποία υπήρχε δημοκρατική ε, λύση το 1960, αλλά τελικώς καταπιέστηκαν από το Νότο και δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν. Ε, πολύ σύντομα θα εκπνεύσουν οι προθεσμίες. Ποια είναι η άποψή σας για την Αφρικανική Ένωση. Τι θα γίνει ε, στη συνέχεια το, στη Σομαλία. Θα ανεξορτατοποιηθεί το Σομαλιλάντ μετά από όλα αυτά. Και μια δεύτερη ερώτηση. Η χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ένωση. Ο κύριο Καντάφη νομίζω ότι κατέβαλε άνω του 20% του προπολογισμού σα. Η νέα κυβέρνηση στην Τρίπολη δεν είναι πολύ ευχαριστημένη παρεπιπτόντω ότι η Αφρικανική Ένωση, ιδιαίτερα τα μεγάλα υποστήριζαν τον Καντάφη στη διάρκεια τη σύγκρουση. Ε, πώς σκοπεύετε λοιπόν να συμπληρώσετε αυτό το κενό στη χρηματοδότησή σα, ε, δεδομένου ότι η Λιβύη δεν θα χρηματοδοτεί πλέον ε, την Αφρικανική Ένωση με την ίδια γεωνοδορία όπω έκανε και στο παρελθόν και τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειακών μπλοκ. Νομίζω ότι η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες οργανώσεις ε, σαν αυτή στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Γκόμες. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς συνεργάζεστε. Υπάρχουν επίσημες ε, συμφωνίες ή συνεργάζεστε απευθείαν με τις κυβερνήσεις χωρίς επίσημη συμφωνία και προσπαθείτε να συντονιστείτε με τις περιφερειακές οργανώσεις. Θα ήθελα να ξέρω πώς λειτουργεί αυτό, διότι δεν έχουμε συγκρίσιμο μέτρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη συνεργάζονται απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν ομάδες περιφερειακών χωρών. Πώς λειτουργεί το σύστημα λοιπόν. Ο κύριο Παντζέρη. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, άκουσα μια περιγραφή των δυσκολιών, των προφανών ε, σειράξεων, κάποιες οι οποίες ε, υφέρπουν και είναι σε αδράνεια, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι σε αντικειμενικά πλαίσια υπάρχει μια δυστοκία. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα με τόση μεγάλη ευκολία. Χωρίς να σταθώ στα προβλήματα στα οποία στάθηκαν και οι συνάδελφοι, να αναφέρω εντάχει τρία. Πρώτον, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα του Σαχέλ θα αποτελέσει θεμελιώδες ζήτημα σε θέματα ασφάλειας και δεν θα αφορά μόνο τις χώρες που εμπλέκονται, ε, κυρίως το Μαλί, αλλά θα αφορά όλη την Αφρικανική Ήπειρο και την Ευρώπη. Ζητώ λοιπόν ε, σε υποστήριξη αυτού του κουαρτέτου, στο οποίο ε, πλήττεται από τη φτώχεια, θα έπρεπε ίσως να προσθέσουμε και το Μαρόκο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ε, εμπλέκεται και το Μαρόκο αλλά θα ήθελα να επαληθεύσετε κατά πόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να υπάρχουν δυνάμεις επιτόπου που ε, προσπαθούν, ε, θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση. Δεύτερον, για το κέρα της Αφρικής. Μόλις αναφερθήκαμε και στη Σομαλία, αλλά εγώ πραγματικά ανησυχώ, διότι ε, υπέρπει μία σύγκρουση ε, στο Τζιμπουτί και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και με την Ερυθρέα, διότι είναι μια κατάσταση η οποία διαονίζεται και θα πρέπει η Αφρικανική Ένωση να πιέσει να βρεθεί μια ισχυρή πολιτική λύση προκειμένου να λυθούν θέματα τα οποία αφορούν την απώλεια οποιοδήποτε δικαίου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει, υπάρχει πλήρης απουσία και ακόμα και μεταναστευτικές ε, κινήσεις προς τη Λιβύη έχουν υπάρξει ακριβώς λόγω του προβλήματος. Τέλος, για τη Δυτική Σαχάρα. Υπάρχει ίσως δυνατότητα να υπάρξει μια στρογγυλή τράπεζα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να υποστηρίζει τη δράση του Κρίστοφερ Ρος. Δεν θεωρώ ότι το να αφήσουμε τα πάντα στα χέρια του υπευθύνου του ΟΗΕ αποτελεί λύση για το πρόβλημα. Θα πρέπει να ε, έχουν και προεξάρχοντα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση για να αποτελέσουν ίσως και ε, κίνητρο για μια πιο καινοτόμο λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου είπατε ξεκάθαρα ότι δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Βέβαια, ήταν τόσο πλούσιες, πλούσιος αυτός ο διάλογος, αυτή, αυτές οι ερωτήσεις, ε, που δυστυχώς πρέπει να τα απαντήσω διαγωνίες και δεν μπορώ να επιστρέψω σε λεπτομέρειες. Ε, πρώτα για τη Δυτική Σαχάρα. Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, εφόσον η τα, σημεία τα οποία θίξατε ε, συνδέονται ουσιαστικά με την ε, ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ε, να δώσουμε νέα όθηση στις προσπάθειές μας για να επιτρέψουμε στον λαό της Δυτικής Σαχάρας να ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση. Η δύσκολη διαδικασία που διεξάγει ο ΙΕ ε, και υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ε, ε, καταδεικνύουν τις δυσκολίες που υπάρχουν, που αντιμετωπίζουμε και που και η Αφρικανική Ένωση αντιμετωπίζει όταν άρχισε να παρακολουθεί αυτή την διαδικασία. Η Αφρική τελικά έδωσε ε, αναγνώρισε ε, το κράτος της ε, Δυτικής Σαχάρας επισήμως. Κατά αυτόν τον τρόπο η Αφρικανική Ένωση αναγνώρισε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας, αλλά και βλέπουμε και την πολιτική βούληση των ε, πολιτικών ηθινόντων που ε, τέθηκαν στη διάθεση του ε, λαού της Δυτικής Σαχάρας. Συμμετέχει λοιπόν πλήρως, με πλήρη δικαιώματα η Δυτική Σαχάρα στην Αφρικανική Ένωση. Η Ένωση εξακολουθεί να θεωρεί ότι υπάρχουν δυσκολίες εφόσον μεγάλο τμήμα δεν βρίσκεται στην, υπό τον έλεγχο του κράτους. Η νευτική διαδικασία λοιπόν συνεχίζεται και δεν μπορούμε να θέσουμε έναν ορίζοντα για την επίλυση του ζητήματο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκέ χώρε επίση έχουν ε, σημαντική ευθύνη για να αξιοποιήσουν την επιρροή του είναι και αυτό ένα σημαντικό ε, στοιχείο για την επίλυση ε, της κρίσης αυτής. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στο λαό της Δυτικής Σαχάρας να εκφραστεί ελεύθερα. Η Άννα Γκόμες έζησε αυτή την κατάσταση ό,τι φορά το Τιμόρ. και όλοι οι λαοί, μεγάλοι ή μικροί, πρέπει να μπορούν να ξεφύγουν από την επικιοκρατία και να ασκήσουν ε, το δικαίωμα της κυριαρχίας τους, που ανοίγει και την προοπτική και για άλλους ε, λαούς στο μέλλον. Για ένα διαφορετικό μέλλον, πιο θετικό. Ίσως η επίλυση του προβλήματος της Δυτικής Σαχάρας ε, να δώσει νέα όθηση και στην δημιουργία του Μεγάλου Μαγκρέμπ. Να δώσω λοιπόν μια δυναμική ολοκλήρωση στην Αφρικανική Ήπειρο. Ε, υπάρχουν πολλές συγκεκριμένε ε, ε, προτάσεις. Νομίζω ότι όλες αυτές οι καλές ιδέες πρέπει να εφαρμοστούν, να ληφθούν υπόψη για να εντοπίσουμε ζητήματα που μας προβληματίζουν αυτή τη στιγμή. Ε, για την, ε, γιατί βεβαίως και ε, παρατηρείται καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυσκολίες στη ζωή των προσφύγων από τη Δυτική Σαχάρα. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε το στομότερο δυνατόν. Γιατί ο λαός αυτός έχει υποφέρει πολύ και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα για την Αφρικανική Ένωση είμαστε σε θέση να δώσουμε, να συνεισφέρουμε στην ε, επίλυση του προβλήματος, πάντα συνεργασία με, τη, με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και με όλους τους άλλους φορείς. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα, στις υπόλοιπες παρατηρήσεις για τις σχέσεις Σουδάν και Νοτίου Σουδάν, όπως ανέφερα, η απόφαση της, ε, ε της της 24 Απριλίου ακολουθήθηκε από, την, ε, από το ψήφισμα 2046 του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας και υπάρχει βεβαίως και καταδικάστηκαν με απόλυτο τρόπο οι βομβαρδισμοί όπως και η εκένωση του Χέγκλη είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο ε, τονίστηκε. Και επαναλαμβάνουμε ότι καταδικάζουμε τους βομβαρδισμούς. Είναι σαφή η θέση της Αφρικανικής Ένωσης. Πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, πρέπει να αποσυρθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις και ο μόνος δρόμος είναι οι διαπραγματεύσεις, ο μόνος τρόπος επίλυσης ε, αυτής της κρίσης. Πρέπει και οι δύο χώρες να κατανοήσουν ότι το πνεύμα και το γράμμα του δικαίου ε, προβλέπει ε, την δημιουργία δύο βιώσιμων κρατών που θα ζουν δίπλα-δίπλα ειρηνικά και το σύνολο της ε, διεθνούς κοινότητας μπορεί να ε, κατευθύνει τις δύο πλευρές ε, για να καταλήξουμε σε μια εξισορροπημένη λύση. Και όπως και να έχει, αυτό είναι προτιμότερο από, από μια κατάσταση σύγκρουσης που έχουμε σήμερα. Για τη Σομαλία. Βεβαίως και Χαιρόμαστε με τις ε, εξελίξεις, ό,τι φορά τη Μισόμ. Έχουμε τη μεγαλύτερη ε, συγκέντρωση σε εκτοπιστέντες στον κόσμο και οι θύνοντες έχουν πάρει όλα τα ε, απαραίτητα μέτρα για να μην υποφέρει ο πληθυσμός. Οι άμαχοι δηλαδή. από αυτές τις ε, στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις. Ε, ο Σαμπάμπ έχει αποσυρθεί, περίπου, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 40 χιλιόμετρα και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. και θα έχουμε νέες θετικές ελεξίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Όπως γνωρίζετε, το στρατηγικό σχέδιο που ανέφερα έχει ήδη εκπονηθεί και και βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο με ε, του ε, υπόλοιπου εταίρου μα, προκειμένου η πολιτική και θεωρητική στρατηγική να οδεύουν χέρι με χέρι. Για να δώσουμε επιτέλους το ένασμα για μια νέα εποχή στην ε, Σομαλία. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτές τις θετικές εξελίξεις για να αποφεληθεί και ο πληθυσμός ε, από αυτές τις νέες θετικές εξελίξεις, από την απελευθέρωση από τον Σαμπάμπ ένα καθεστώς ε, αρκετά σκληρό που επέβαλε ιδιαίτερα κατακριτές ε, πρακτικές. Σε ό,τι αφορά το Μαλί και την Κινέα Μπισάου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ευθυγραμμιζόμαστε απολύτως ε, με τα όσα είπατε ότι αυτές οι αρνητικέ εξελίξεις που βλέπουμε έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού. Ε, όλα τα πραξικοπήματα είναι αρνητικά, ιδιαίτερα αυτά στο Μαλί και στην ε, και στις δύο περιπτώσεις ε, βρισκόμαστε στη διαδικασία ε, εκλογών. Έτσι έχουμε επικίνδυνη υποχώρηση στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της ε, Αφρικής και είναι απαραίτητο να μεριμνήσουμε ούτω ώστε να μην ε, ε, επιτρέπουμε την διάπραξη προξικοπημάτων. Η καταδίκαση τέτοιων ε, κινήσεων από τη διεθνή κοινότητα είναι ο μόνος ε, δυνατός ε, τρόπος με σεβασμό των κύριων θέσεων που έχουν εκφραστεί και βεβαίως με το να συγκεντρώσουμε το σύνολο των φορέων για την επίλυση της κρίσης. Και ήδη για τις 7 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί μια συνεδρίαση ε, ε στήριξης και παρακολούθησης ε, της ε, Σομαλίας, στην οποία συμμετέχουν και διεθνείς εταίροι σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένα Έθνη και άλλοι φορεί ε, και το απόγευμα τη ίδια ημέρα θα έχουμε μια διεθνή ομάδα επαφής για την Γουινέα Μπισάου με την οποία θα συμπροεδρεύσει και η ΣΕΛΕΠΕ και η ΣΕΝΤΕΟ. Στις 7 Ιουνίου ελπίζουμε λοιπόν ότι η Αφρικανική Ένωση θα βγει πιο ισχυρή και θα εκφράσει με ακόμα πιο ξεκάθαρο τρόπο την βούλησή της να εργαστεί και σε αυτό το πεδίο, στο Μαλί και στην Κουιναμπισάου. Για τον Νταρφούρ, ναι πράγματι έχει μειωθεί η ανασφάλεια ε, και η έλλειψη σταθερότητας ε, ε, σε αυτή την περιοχή. Μας αφορούν κυρίως το, το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν αυτό το πρόβλημα, αλλά βεβαίως και το Νταρφούρ είναι μια ζώνη κινδύνου εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι ε, οπλισμένες ομάδες που δεν έχουν υιοθετήσει το έγγραφο που υιοθετήθηκε στην Ντόχα. από τον ε, αρμόδιο διαμεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών. Επομένω, ε, θα πρέπει να επιλύσουμε και τις υπόλοιπες ε, ένοπλες ομάδες να προσυπογράψουν το κείμενο της Δόχα. και να ληφθούν υπόψη και ε, τα αιτήματα ενδεχομένω και αυτών των ε, δυνάμεων. Όμως οι στρατιωτικές επεμβάσει δεν είναι επιλογή. Και αυτό θα πρέπει να το καταστήσει σαφές ε, και η διεθνής κοινότητα. Αναφέρθηκα στην εξέλιξη αυτό το συγκρούσεων και σας είπα ότι όλες αυτές οι συγκρούσεις ε, ε, διεξάγονται σε εσωτερικό επίπεδο, στο πλαίσιο ενός ε, κράτους και όχι σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για ένοπλες συγκρούσεις σε εσωτερικό επίπεδο. Εντό των εσωτερικών συνόρων, λοιπόν, αλλά πολλέ φορέ υπάρχουν και άλλοι φορεί που επεμβαίνουν έξω από τα σύνορα αυτή τη χώρα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτές είναι επιχειρήσεις, ε, ε, είναι τρομοκράτες, ε, πειρατές. Θα μπορούσαμε σε πολιτικό επίπεδο να δώσουμε και μια τέτοια ανάλυση. Και εγώ δεν, προσωπικά δεν είμαι αντίθετο, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε για την ενίσχυση της ε, διεθνούς δράσης στο Μαλί και το Βόρειο Μαλί. Αναφερθήκατε στις ε, δηλώσει του Γάλλου Προέδρου. Χαιρόμαστε που ε, κινητοποιείτε σε αυτόν τον τομέα. Θα θέλαμε το σύνολο της διεθνούς κοινότητας στεναρά να απορρίψει τον κατακαιρματισμό. Η Αφρική θα πρέπει να οδεύσει προς ε, την ολοκλήρωση μέσω του διαλόγου όταν αυτό αρκεί ε, και με την προσφυγή σε άλλα μέσα, ενδεχομένως και ε, στρατιωτικών δράσεων, ενεργειών, όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο. στο πλαίσιο των δημοκρατικών ε, θεσμών ε, που έχει κατακτήσει το Μαλί εδώ και 20 χρόνια ε, υπάρχει δυνατότητα όλες οι κοινωνικές διαστρωματώσεις να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να χρειάζεται να εξεγερθούν, να πάρουν τα όπλα και να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία του, της χώρας. το πραξικόπημα αυτό αποδυνάμωσε το Μαλί γιατί έτσι έχασε το μεγαλύτερο ε, όπλο του το Μαλί που ήταν ε, η νομιμότητα. Στο βόρειο Μαλί ε, πρέπει ω διεθνή κοινότητα να ενθαρρύνουμε τον ε, διάλογο για την ε, εξέβρεση μια ειρηνική ε, λύση στα προβλήματα των Τουαρέγ, τα οποία συνδέονται με την νομιμότητα τη εθνική κυριαρχία του Μαλή. Και βεβαίως να είμαστε πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διεθνούς ε, Τρομοκρατία, Να μην επιτρέψουμε στη διεθνή τρομοκρατία να κερδίσει έδαφος ε, και να ε, επεκτείνει την επιρροή της στα δύο τρίτα της επικράτειας του, του, νόριου, του Βόρειου Μαλή που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Τώρα, για τη χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ένωσης δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο από ότι ο κ. Γκαντάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα εδώ, επομένω δεν έχουμε ουσιαστικά προβλήματα. Αλλά πιο σοβαρά να σα απαντήσω ότι ο Γκαντάφη δεν πλήρωσε ποτέ το 20%. Η μεγαλύτερη ε, συνεισφορά πέντε ε, κρατών μελών ε, που πλήρωναν επίση όρη ήταν πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων ε, Λιβύη και άλλοι. Και έτσι φτάνουμε στο 12-13%. Επομένω, ποτέ ο Γκαντάφη δεν συμμετείχε σε μεγαλύτερο βαθμό στην χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ένωσης. Η Αφρικανική Ένωση πάντα βασίζεται στην, ε, στη χρηματοδότηση από όλα τα κράτη-μέλη και, και σε αυτά τα πέντε κρατημέλη που σας ανέφερα, αλλά και ε, στους διεθνείς ε, εταίρους. Σκεφτήκαμε και άλλα μέτρα, όπως ε, την ε, αύξηση των συνεισφορών, και θεωρούμε ότι υπάρχει κίνητρο για τα κράτη-μέλη μας να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό για να μειώσουμε το μερίδιο που επομίζονται οι υπόλοιποι εταίροι μας. Ε, το νέο ε, καθεστώς της Λιβύης έχει πληρώσει, έχει εξοφλήσει τις, ε, το μεριδιό του. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Βεβαίως ο καιρός περνάει γρήγορα δεν έχω πολύ χρόνο. Κλείνοντα, ε, να πω ότι σε ό,τι αφορά την ε, σύνδεση μεταξύ της, ε, της Αφρικανικής Ένωσης και της Περιφερειακής Επιτροπής, υπάρχει η αρχή της επικουρικότητα. Υπάρχει αρχή επιμερισμού των, ε, των ε, ευθυνών ε, και του άχθους, αρχής συμπληρωματικότητας των προσπαθειών, η Επιτροπή των Περιφερειακών Οργανώσεων είναι αναπόσπαστο τμήμα της όλης αυτής της διαδικασίας. Από αυτή την πλευρά λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει βεβαίως να εμπνευστούμε από το ευρωπαϊκό παράδειγμα και να ε, αναπτύξουμε τις δικές μας ε, βέλτιστες πρακτικές και όπως σας είπα προηγουμένως ελπίζουμε το 2013 που θα είναι που θα στην την 50η επέτειο από την έναρξη της Αφρικανικής, ε, Αφρικανικής Ένωσης θα δώσει μια νέα όθηση στον Παναφρικανισμό και θα συμβάλλουμε περαιτέρω ε, στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και στην ολοκλήρωση των εταιρικών μας σχέσεων με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε και νομίζω ότι ήταν και ιδιαίτερα χρήσιμη και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι ότι καλύτερο.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 Meine Damen Κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά να καλωσορίσω εδώ ανάμεσά μας τον πρόεδρο της ΕΟΚΕ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Κοινότητας, καθώς επίσης και την κυρία Γκράμπε, διευθύντρια του Open Society Institute των Βρυξελών, την οποία γνωρίζετε όμως από την προηγούμενη ιδιότητά της. Ε, και σήμερα θα κάνουμε μια κοινή συζήτηση για τη διεύρυνση, τα πολιτικά ε, κριτήρια και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Η έκθεση της κυρίας Κοπά κατά την άποψή μου θα αποτελέσει ορόσημο για το μέλλον και θεωρώ ότι θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και με αποτελεσματικό τρόπο. Σήμερα γίνεται η δεύτερη συζήτηση για την έκθεση της κυρίας Κοπά και η συνέχεια αυτής της συζήτησης θεωρώ ότι επιβάλλεται ο κύριος Νίλσεν και η κυρία Γκράμπε είναι δύο εκπρόσωποι γνωσμένου κύρους που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να προσφέρουν σε αυτή τη συζήτηση και θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Θα δώσω λοιπόν στον καθένα από εσά από 5 έως 10 λεπτά. Ε, να σας πω ότι ε, έχετε προνόμια σήμερα, διότι στους ευρωβουλευτές ένα-δύο λεπτά θα δώσουμε. Κύριε Νίλσεν, έχετε το λόγο. thank you very much, Brook, for... Ευχαριστώ πολύ για την ε, ευκαιρία αυτή. Θα ευχαριστήσω επίση την εισηγήτρια, την κυρία Κοπάη, ε, το προσχέδιο έκθεση της, το, την οποία τη διάβασα και νομίζω ότι συμφωνώ σχεδόν με όλα τα 22 σημεία τα οποία περιλαμβάνει. Ε, δίδεται στην έκθεση έμφαση στις δίκες συνθήκες για τις υποένταξη χώρες. Και σίγουρα το υποστηρίζω από την πρώτη μέρα πρέπει και οι πολίτες και οι πολιτικοί τους να γνωρίζουν το ποιος είναι ο δρόμος εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αυτό καθιστά πιο απλό για τους ε, πολίτες των υποένταξη χωρών να αξιολογούν την, το έργο των πολιτικών τους. Αυτό όμως Σημαίνει επίσης ότι και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι δίκαια και να τηρούν τις ε, δεσμεύσεις τους. Acta sum servanta, όπως λέμε στα λατινικά. Ε, βέβαια υπάρχουν ε, ε, ε όροι για την ένταξη και είναι γνωστή ποιοι είναι αυτοί οι όροι, αλλά κάθε διαδικασία ένταξης είναι μια διαδικασία μάθησης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις εμπειρίες προηγούμενων εντάξεων θα πρέπει να διδασκόμαστε και να προσαρμόζουμε την ε, τακτική μας. Θα πάω κατευθείαν στα σχόλια της ΕΟΚΕ. Πού πιστεύουμε δηλαδή ότι θα πρέπει εμείς να συνεισφέρουμε. Ε, Θέλουμε η, ε, ε, θέλουμε η, η διαδικασία διεύρυνσης να ε, μην είναι οδυνηρό, να μην είναι κάτι οδυνηρό, δηλαδή μείωση της ανταγωνιστικότητας, οι κίνδυνοι για την οικοδομία, όπω πολλέ φορέ το δέχονται, το, αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Οι κοινωνικέ πολιτικέ θα πρέπει να λάβουν ιδιαίτερο βάρο. και θα πρέπει να ενημερώνουμε του πολίτε, Για παράδειγμα, το κοινωνικό κεκτημένο για την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασία. ο, το μέγιστο αριθμός ωρών εργασίας ανά ημέρα, όλα αυτά είναι επιτυχίε Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του κοινωνικού κεκτημένου. Η πρόταση τη ΕΟ και γι' αυτό το σημείο, την κοινωνική διάσταση δηλαδή, ε, έχει επίσης ε, σχέση και με τον κοινωνικό διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να τονιστεί. Το λέτε στο σημείο 9 της έκθεσης. Θέλουμε ε, ο κοινωνικός διάλογος να προωθηθεί στις ένταξη χώρες, γιατί έτσι η ενταξιακή διαδικασία θα είναι πιο ενδιαφέρουσα για αυτές τις χώρες. Η διεύρυνση δεν πρέπει να είναι μόνο στα χέρια της, δημο, της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης. Είναι και θέμα πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες, αλλά και το θέμα κοινωνικών εταίρων και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως επίσης αναφέρεται. Θα πρέπει όλοι αυτοί να συμμετάσχουν, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να γίνει επιτυχώς αυτή η διαδικασία. Για την κοινωνική διάσταση να πω και το εξής. Σε όλες τις υποένταξη χώρες χρειάζεται ισχυρότερη παρουσία των συνδικάτων. Η, ε, τα συνδικάτα σημαίνουν, σημαίνουν, σημαίνουν επίσης και ισχυρές εργοδοτικές οργανώσεις. Ε, τα ε, συνδικάτα των όμως έχουν ιδιαίτερο ρόλο να παίξουν στην προσαρμογή της χώρας, της κάθε χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει περισσότερη βοήθεια προς τα συνδικάτα για να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και στους κοινωνικούς, ε, οι κοινωνικοί εταίροι και ιδιαίτερως στα συνδικάτα θα χρειάζονται τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμμετάσχουν επιτυχώς στις διμερείς και τριμερείς κοινωνικούς διαλόγους. Ασφαλώς και θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα συνδικάτα αντιπροσωπεύουν πραγματικά τους εργαζόμενους και ότι είναι ανεξάρτητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της διάβνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπογραμμίσω το εξής. Ε, είναι πραγματική πρόκληση ε, να πείσουμε τους πολίτες σήμερα. Να τους πείσουμε δηλαδή ότι η διεύρυνση θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα. Όμως μην ξεχνάμε ότι οι προσδοκίες είναι τεράστιες στον πληθυσμό των υποένταξη χωρών. Και θα πρέπει κάθε ένταξη να θεωρείται ως ιστορική ευκαιρία για την Ευρώπη να ενωθεί. Υπό την προπόθεση βέβαια ότι οι υποένταξη χώρες πληρούν τα κριτήρια. Πιστεύω όμως ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγματι ιστορική πρόκληση να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί. Θα, ε, εμείς στην Επιτροπή μας χρησιμοποιούμε κυρίως δύο εργαλεία. Πρώτον, έχουμε δημιουργήσει την, τι, κοινέ ε, συμβουλευτικές επιτροπές για κάθε μία από αυτές τις υποένταξη χώρες. Ε, ε, με βάση τις συμφωνίες σταθερότητας και γνωρίζω ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως θα είχαμε τη δυνατότητα στο μέλλον να συνδιοργανώνουμε συναντήσεις ε, Δηλαδή όταν εσείς ε, συναντάτε τους πολιτικούς, εμείς την ίδια μέρα να συναντούμε τους κοινωνικούς εταίρους από αυτές τις χώρες. Μετά, έχουμε, ε, έχουμε το φόρμ της κοινωνίας των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα, ε, μια εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια με, τις, με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών της συγκεκριμένη περιοχής. Φέτος θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου το τέταρτο τέτοιο φόρουμ και ε, αντιμετωπίζουμε ανησυχίες όπως αυτές που έχετε εσείς ε, στην έκθεση ε, ανεργία, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης κλπ. Ορισμένες από τις συστάσεις μας θα αποσταλούν στους πολιτικούς ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια. Θα, μετά θα εργαστούμε για την υλοποίησή τους μαζί με τους εταίρους μας, τους κοινωνικούς μας εταίρους στην περιοχή. Τελειώνοντας, να πω το εξή. Η ΕΟΚΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει την συνέχιση της διεύρυνσης. Είναι μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χάσουμε. Όμως θέλουμε η διαδικασία αυτή να είναι δικαίη, ε, να μην αποκλείει κανέναν ε, και να είναι διαφανής. Θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα καλύτερο βαθμό προετοιμασία σε αυτές τις χώρες πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί όμω στενά με την κοινωνία των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία. Εμεί εργαζόμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ελπίζω ότι θα μα υποστηρίξετε και εσεί. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας μιλήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριε Γκρέβερ. Και εγώ έχω εργαστεί για τη διεύρυνση εδώ και 20 χρόνια στην Κομισιόν και ως ακαδημαϊκός, σε think tanks κλπ. Σήμερα εκπροσωπώ την Open Society Foundations ε, Νομίζω ότι η διεύρυνση αφορά και τις χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, τις χώρες των Βαλκανίων και της Τουρκίας και την Τουρκία. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κοπά για την έκθεσή της ε, που υπογραμμίζει πολλά πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Ε, εμείς εργαζόμαστε εδώ και 30 χρόνια σε χώρες υποδιεύρυνση ε, και στις χώρες που ακόμα δεν έχουν γίνει μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, συμπίπτουν τα συμπεράσματά μας ιδιαίτερο στο σημείο F για την δίκαιη και διαφανή αξιολόγηση. Επίσης τη χρήση των benchmarks που είναι πολύ σημαντικά για την αξιολόγηση πρόοδου αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργούν πρόσθετες, πρόσθετους όρους που δεν ήταν μεταξύ των αρχικών όρων. Επίσης το σημείο 20. Η πρόταση τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να αξιολογούνται σε ό,τι αφορά την προσήλωσή τους στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ε, πρέπει να ισχύουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για τις παλιές και τις κοινωνικές χώρες. Γιατί η πολιτική εξέλιξη μιας ε, χώρας ε, η ποιότητα της δημοκρατία της ε, δεν ε, τελειώνουν τη στιγμή που θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη δεν είναι το τέλος του ταξιδιού. Γιατί το να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη οικογένεια αρχών. Η θα πρέπει όμως να ελέγχεται το κατά πόσον τηρούνται αυτές οι αρχές. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι είδους ε, μηχανισμό θα μπορούσε να δημιουργηθεί για την παρακολούθηση αυτή. Το άρθρο 7 και το άρθρο 258 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν δίνουν πολλές λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά την διεύρυνση, το σημαντικό είναι να ε, τονίσουμε την ανάγκη λογικής συνέπειας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών προτύπων και απαιτήσεων. Δηλαδή τα νέα κράτη-μέλη ε, δεν θα πρέπει να ε, κρίνονται με βάση χειρότερα, πιο αυστηρά στάνταρ. Θα πρέπει όλες οι χώρες, και οι καινούς και οι παλιές, ε, να τίνουν, να βελτιώσουν την ποιότητά τους. Ε, να μην περιοριζόμαστε δηλαδή μόνο στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Πρέπει το Κοινοβούλιο ενδεχομένω να εξετάσει ποιο θα πρέπει να είναι αυτό ο μέγιστο κοινό παρανομαστή σε διάφορα θέματα όπω ε, θεμελιώδη δικαιώματα ε, και άλλου είδου δεσμεύσει των κρατών μελών. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που έχω σε θέματα διεύρυνση Το Open Society Foundation και, στην, και στην Κομισιόν είναι ότι ε, ε, η, είναι πολύ σημαντική η ικανότητα των θεσμών και των θεσμικών οργάνων του κάθε υποένταξη κράτους να εφαρμόσει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όπως περιγράφονται στα κριτήρια της Κοπενχάγης. Συνεπώς, η θεσμική ικανότητα της κάθε χώρας είναι πολύ σημαντική και η σταθερότητά τους. Έτσι, η σταθερότητα και ποιότητα των θεσμών και των θεσμικών ικανοτήτων. Αν δηλαδή μπορούν τα όργανα να λειτουργήσουν, τότε θα λειτουργήσει και η χώρα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρεις παρατηρήσεις από την, από την εμπειρία των Open Society Foundations, ε, ιδιαίτερος για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό η κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει και θα την όριζα την κοινωνία των πολιτών ως ένα πλατή φάσμα ε, οργανώσεων της κοινωνίας στην, κάθε χώρα. Ε, εργοδότες, ε, συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μικρές τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, σωματεία, ενώσεις, όμιλοι επιχειρήσεων, ε, ένα μεγάλο φάσμα οργανώσεων τα οποία αποτελούν ε, την ε, κοινωνία των πολιτών. Μέχρι τώρα η Κομισιόν έχει πλησιάσει αυτές τις ομάδες μέσω του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών που έχει λάβει διάφορες μορφές. Αυτό που είναι όμως ζωτική σημασία είναι η προσέγγιση αυτή να συνδέεται με δύο πράγματα στα οποία ο ρόλο του Κοινοβουλίου είναι σημαντικό. Πρώτον, ε, συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλέ επαφέ προφανώ, αλλά τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά προκειμένου τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με την κοινωνία των πολιτών, την τοπική κοινωνία των πολιτών. Δεν πρέπει η ενταξιακή διαδικασία να είναι απλώ μια πολιτική ε, συνεργασία, μια πολιτική διαβούλευση ανάμεσα σε την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το Εθνικό Κοινοβούλιο της υποένταξη χώρας να μην λαμβάνει μέρος. Και ταυτόχρονα το Εθνικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Συνεπώς ε, η, ε, δεν θα πρέπει η διαδικασία ένταξης να αποκοπεί από την κοινωνία των πολιτών. Δεύτερο σημείο, κάτι το οποίο το λέει η έκθεση, είναι η σημασία ε, ε σαφούς και σταθερής πολιτικής από της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τόσο από πλευρά κρατών μελών όσο και από πλευρά των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει όλα να είναι ε, προσιλωμένα στην ένταξη. Αυτό είναι δύσκολο και είναι δύσκολο ε, σε μια υποένταξη χώρα να διατηρηθεί η μεταρρυθμιστική ορμή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθαρή. Θέλουμε ή δεν θέλουμε αυτή τη χώρα. υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο πρώτος κίνδυνος ε, είναι ε, το ζεστό κρύο, μια συνεχής αναλλαγή ζεστού κρύου σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την υποένταξη χώρα. Ε, ταυτόχρονα όμως είναι εξίσου επικίνδυνο το εξής. Επειδή ορισμένες χώρες είναι ε, να θεωρείται ότι επειδή η ε, έναξη χώρα έχει συγκεκριμένους φίλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ιστορική φιλία με συγκεκριμένες χώρε, να μην χρειάζεται, να θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να πληρεί τα κριτήρια. Και οι δύο αυτοί οι είναι σημαντική. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρεί τις δεσμεύσει τη, 20 χρόνια μετά την, ε, τον καθορισμό των κριτήριων τη Κοπεχάγης ε, αυτά τα κριτήρια ε, έχουν δείξει την ανάγκη, την αξία του. δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, μειονότητε, ε, κράτος δικαίου όλα αυτά είναι πραγματικά κριτήρια τα οποία είναι επίκαιρα και, σήμερα. και σήμερα θα πρέπει να δούμε την οικονομία τη αγορά, την ανταγωνιστικότητα, όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα ιδιαίτερα με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στα Βαλκάνια και από πολιτιστική και από οικονομικής πλευράς ε, ε, χρειάζεται οι μεταρρύθμιση να ξεκινήσουν νωρίς και να παρακολουθούνται ιδιαίτερα στο δικαστικό στη δικαστική εξουσία γιατί η ποιότητα των θεσμών είναι ιδιαίτερα σημαντική για να εξασφαλιστεί η συνεχής η συνέχιση της πορείας μετά την ένταξη. Ε, χρειάζεται ένα πολιτιστικό ήθος σε ό,τι αφορά την ε, τη λειτουργία της δημοκρατίας και θα πρέπει τα θεσμικά όργανα σε εθνικό επίπεδο ε, να είναι συνδεδεμένα με την κοινωνία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Να σας υπενθυμίσω γιατί βλέπω ότι πολλοί από εσά έχουν εργαστεί σε θέματα διάμεση για πολλά χρόνια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλη η κοινωνία συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία. Το μόνο που δεν είδα στην έκθεση είναι ε, ότι και οι πιο ευάλωτοι, τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού θα πρέπει να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, η Ρωμά. Σε πολλά κράτη-μέλη και σε πολλά υποένταξη κράτη υπάρχουν Ρωμά οι οποίοι είναι εκτός διαδικασίας. Γι' αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν ε, εθνικές διαδικασίες ένταξης οι οποίες δεν θα χρειαζόντουσαν αν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ένταξης ε, από τη δεκαετία του 70 και μετά είχε ληφθεί ήδη υπόψη η κατάσταση των ευάλωτων κομματιών για παράδειγμα τον Ρώμα η Ρωμά είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση αυτή τη κοινωνική διάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. για την παρουσίασή σας. Τώρα, συνάδελφοι, θα ήθελα να καλέσω την εισηγήτρια να πάρει το λόγο αρκετά σύντομα για να συνεχίσει και η συζήτηση. Thank you, Chairman. Uh, first of all... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΑΦΕΤ και εσά, ε, Πρόεδρε, προσωπικά για την δεύτερη δυνατότητα που μου δίνετε για να συζητήσουμε ε, αυτό το ζήτημα τη διεύρυνση μετά και τις δύο πολύ ενδιαφέρουσες ε, ε, επεμβάσεις, ε, εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην διαδικασία. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Νίλσεν που αποδέχθηκε την θέση μας για την ε, θέση της ΕΟΚΕ στο ζήτημα. Ξέρουμε ότι η Επιτροπή έχει ως στόχο την ενίσχυση της ε, νομιμότητας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δίνοντας δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να εκφράσει τις απόψεις της ευρωπαϊκού επίπεδο. Ε, θεωρούμε ότι είναι φυσικό ε, εταίρος μας λοιπόν σε ό,τι αφορά την διεύρυνση. Γι' αυτό θέλω να υποβάλω τροπολογία που θα τονίζει τον ε, ρόλο τη και θα καλεί για ενίσχυση της συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημείωσα δύο πολύ σημαντικά σημεία που αναφέρατε, Πρόεδρε, για την ανάγκη ενίσχυσης των σωματείων αλλά και την ε, ανάγκη ε, στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε για το κοινωνικό φόρουμ. Εδώ να ευχαριστήσω και την ε, Heather Grab, που ασχολείται με ζητήματα διεύρυνσης εδώ και πολλά χρόνια. και στο κείμενό τη βλέπουμε και μια πιο ακαδημαϊκή ανάλυση του ζητήματος. Έχω ένα τεχνικό ερώτημα ε, για την κυρία Γκράμπερ που συνδέεται με την ε, ε, εποπτεία της διαδικασία διεύρυνση. Στην έκθεσή μου χαιρετίζω την πρόθεση της Επιτροπής να θέσει benchmarks, να θέσει κάποια σημεία, κάποιους δείκτε που πρέπει να τεθούν σε όλε τι διαδικασίε, σε τι φάσει φάσεις διαδικασίας, όχι μόνο στι διαπραγματεύσεις, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η διαφάνεια τη όλη ε, όλης διαδικασίας. Ε, από την πείρα σα θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό από πρακτική άποψη. Θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό που είπατε στο ίδιο μικρό των τον κύριο για την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και θεωρώ πολύ σοβαρό την, σημείο την συμμετοχή των ευαίσθητων πολιτικών ομάδων, θα προσπαθήσω, ε, κοινωνικών ομάδων, θα προσπαθήσω να το θίξω και στις τροπολογίες και να το διορθώσω. Ε, αναφέρθηκα σε έναν ε, μηχανισμό παρακολούθησης υποπτίας στα υφιστάμενα κρατημέλη για να ελέγξουμε την συμμόρφωση με τους όρους της Κοπεχάγης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά που πλήττουν την αξιοπιστία μας. Ε, με καθησυχάζει λοιπόν το γεγονό ότι θεωρείται ότι είναι καλή ιδέα. Βεβαίως πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Όμως έτσι μπορούμε να σταματήσουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, και όπως είπατε, η προσχώρηση, η ένταξη δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Η διαδικασία συνεχίζεται και μετά πώς μπορούμε να πετούμε τη συμμόρφωση από άλλους ε, όταν και εμείς οι ίδιοι δεν ε, ε, ακολουθούμε πλήρως τις ίδιες προϋποθέσεις για τα κριτήρια. Σας ευχαριστώ και πάλι και περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Κοπά αλλά και τους ε, δύο εμπειρογνώμονε που ε, μα έκαναν τι παρουσιάσει. Είπατε ότι πρέπει να είμαστε σύντομοι. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω λοιπόν αρχικά. Είναι μια πολύ καλή έκθεση. Σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ με τα όσα αναφέρει η κυρία Κοπά. Όμως, Πρόεδρε, θεωρώ ότι σε ορισμένα σημεία θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία. Στην έκθεση, κυρία Κοπά κάτι το οποίο λέει εδώ και πολλέ πολλές φορές, μιλάει για τα, για τα διμερεί ζητήματα, τα οποία δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για την διαδικασία προσχώρηση. Ένταξη. Αυτό τι σημαίνει όμως ακριβώς, ότι ε, τα αφήνουμε να συνεχίσουν ή ότι πρώτα υπάρχουν διαβουλεύσεις για να απευθυνθούμε μετά στο, ε, ε, στο δικαστήριο για να επιληθεί εκεί η διαδικασία. Γιατί νομίζω ότι σε αυτήν την περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Πρόεδρε, θεωρώ ότι δεν είναι σαφές το εξή. Παράγραφος 6. Η ε, κυρία Κοπά μιλά για, την ικανότητα ενσωμάτωσης, αλλά αυτό θα πρέπει να εκαταστεί σαφέστερο, Πρόεδρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν τέτοια δικαιοσύνη, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να, να, να είναι κύριε προτεραιότητε η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό πρέπει να αναφέρεται ω σαφή προτεραιότητα. Μετά, για την κοινωνική πτυχή, η κυρία Κοπά τονίζει και ε, αυτέ τι πτυχέ. Ε, συμφωνώ μαζί τη λοιπόν προ αυτό. Όμω, έχω το εξή ερώτημα. Θα θέσουμε μπορούμε να αναπτύξουμε ένα τέτοιο σύνολο κοινωνικών κριτηρίων. Δεν ισχύει ότι με τα υφιστάμενα κριτήρια υπάρχει ήδη περιθώριο για τα κάτι μελη ε, όχι μόνο να τα, να τα κατηγορήσουμε, να τα καταδικάσουμε, αλλά και να τα στηρίξουμε. Κάτι άλλο το οποίο θεωρώ ε, σημαντικό είναι η γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής Προπολογισμού. Εκεί αναφέρεται ότι το υποψήφιο κράτο μέλο πρέπει να λάβει μεγαλύτερη στήριξη για να ε, συμμορφωθεί με την ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ. Άλλο σημείο. Ε, τι συμβαίνει με τα υφιστάμενα κράτη-μέλη. Και, για αυτά τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια δεν πρέπει να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο εδώ. Αυτά είναι, συντομία, τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Κύριε Κορνέλισεν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σχόλια του κύριου Νίλσεν και συμφωνώ απολύτως με τις ανησυχία του ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές πτυχές στη διαδικασία της διεύρυνθης. Εγώ ήμουν συντάκτηρα της γνωμοδότησης ε, για το EPA2 και τα θέματα τα οποία αναφέρεται είναι αυτά τα οποία προσπάθησα να αντιμετωπίσω και εγώ στην γνωμοδότησή μου. Ότι πρέπει να ενισχύσουμε του κοινωνικού εταίρου και τον κοινωνικό διάλογο πολύ περισσότερο. Ότι είναι κάτι εκ διαμέτρου αντίθετο με την υπόλοιπη κοινωνία των πολιτών. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν νομοθετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω, εάν οι χώρε προ προσχώρηση θέλουν να συμμετέχουν πλήρω σε αυτό στο μέλλον, θα πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερη προσοχή στο σημείο αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την εφαρμογή του κοινωνικού κεκτημένου. Υπάρχουν βεβαίως ε, ε, ένα ιδιαίτερο αμάλγαμα ε, θεμάτων που είναι ήδη εφαρμοσμένα. Υπάρχουν θέματα επιθεωρήσεων εργασίας, ε, το μη ε, ε, εργαζόμενοι οι οποίοι δεν δηλώνονται και όλα αυτά είναι τμήμα της διαδικασίας διεύρυνσης και θεωρώ ότι είναι λυπηρό ότι μας απασχολούν πολύ περισσότερο πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά αλλά τα κοινωνικά ζητήματα και τα εργασιακά ζητήματα είναι θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινότητας των πολιτών. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι η κυρία Κοπά αναφέρει πολλά από τα ε, σημαντικά σημεία ε, που μας απασχολούν το γεγονός ότι υπάρχει ε, πολύ μεγάλη επιρροή σε εκλογικά θέματα στα κρατη ε, όχι τόσο στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο Συμβούλιο Υπουργών. Εκεί ε, το τι γίνεται σε εκλογικό επίπεδο για τους διάφορους υπουργούς φαίνεται ότι διαδραματίζουν έναν αδικαιολόγητο ρόλο για τους υπουργούς, ενώ δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει τόσο στην πρόοδο που έχουν επιτύχει οι χώρες οι οποίες θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα, για κάποια θέματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να επιληθούν, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της διεύρυνσης και θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο για να διευθετούμε αυτά τα ζητήματα, ε, να τα αντιμετωπίζουμε κάπου αλλού, ώστε να μην δηλητηριάζουν την αξιοπιστία και τη συνέπεια της διαδικασίας της διεύρυνσης. Η κυρία Κοπά αναφέρεται σε πολλά από αυτά τα στοιχεία. Κατά πάσα πιθανότητα θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσουμε το χαρακτήρα της έκθεσης. Ίσως θα συμπεριλάβουμε και κάποια από τα κοινωνικά ζητήματα ζητήματα τα οποία αναφέρθησαν και είμαι βέβαιη ότι τελικώ θα καταλήξουμε σε ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοπά, θέλετε να απαντήσετε στους συναδέλφους. Ναι. Μόνο κάτι να πω για τα διμερεί ζητήματα. Ζήσαμε όλοι την αντίθεση μεταξύ της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να αποτελούν πρόσκομα στη διεύρυνση και την της πραγματικότητας. Το σκεπτικό μου ήταν να υπάρχει μια διατύπωση που μπορεί να συνδυάσει την πραγματικότητα με τη βούληση του Κοινοβουλίου. Όπερ και ότι θα πρέπει να επιλύονται σε διαφορετικά φόρουμ και ε, έδωσα κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί να επιληθούν μέσω διεθνούς δικαστηρίου, μέσω διατησίας, ε, μέσω ε, εμπλοκής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην δηλητηριάζουν την όλη διαδικασία και να μην τα αφήνουμε να ε, ε, σέρνονται στην όλη διαδικασία εντό εισαγωγικών διότι ε, αποτελεί γεγονό ότι στο Συμβούλιο μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ω εμπόδιο να πάσα στιγμή. Ό,τι και να πούμε εμεί, ό,τι και να πει μια κυβέρνηση, δεν είναι ωραίο να έχουμε μια εντελώ αντίθετη θέση από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Γκράμπε. Να αναφερθώ και εγώ στο ερώτημα που έθεσε η κυρία Κοπά για το benchmarking. Νομίζω ότι αυτό σχετίζεται και με τα θέματα των διμερών θεμάτων που μόλι αναφέρατε. Διότι όπω είπατε κι εσεί, ανα πάσα στιγμή μπορεί κάποιο να θίξει το θέμα του ε, διμερούς προβλήματος. Ενώ το benchmarking είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητηθούν ζητήματα που δεν έχουν τόση σχέση με τα κριτήρια τη Κοπενχάγη, αλλά με διμερή προβλήματα. Και νομίζω ότι σε κάθε στάδιο θα πρέπει να δούμε σε τι με τι θα σχετίσουμε τα διάφορα ορόσημα. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή εφαρμόζει συγκεκριμένα ορόσημα για κάθε ε, καθεστώ, παραδείγματο χάρη για το καθεστώ τη υποψήφια χώρα. Δεν τα είχαμε για τις χώρες οι οποίες εντάχθηκαν το 2004 και το 2007, αλλά πλέον είναι ένα απόσπαστο τμήμα της διαδικασία. Στο δρόμο λοιπόν προς την ένταξη είναι πολύ σημαντικά, διότι ο δρόμος για την Τουρκία και τα Βαλκάνια είναι πολύ μακρύς και θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κάποια σημεία που θα τους ενθαρρύνουν στη διάρκεια της διαδρομής και είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε και τη μόχλευση που παίρνουμε από αυτά ώστε να βοηθήσουμε τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στις χώρες ε, επιβραβεύοντας την πρόοδα, δίνοντας κίνητρο ή και για να μπορέσουμε να πούμε σε μια χώρα ότι δεν κάνετε αρκετά, για παράδειγμα για τα δικαστικά ζητήματα ε, ή κάποια άλλα που μπορεί να έχουν σημασία σημασία για την πρόοδό Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνεται διαχωρισμό των διαφερών φάσεων και να δημιουργούνται κίνητρα ώστε να προχωρά κάποιο. Για τα ορόσημα λοιπόν αυτά, θα θέλαμε να έχουμε και κάποιες ε, προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται. Μόλι φτάνει κάποιο λοιπόν σε κάποιο benchmark, σε κάποιο ορόσημο, ε, το Συμβούλιο θα θέλει να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό είναι ότι προσθέτουμε και άλλα διμερεί ζητήματα στη διαδικασία. Αν είναι προδιαγραφέ, standards, θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιείται αυτό ο όρο κατά με, διότι μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες δεσμεύσει που ανέλαβε μία χώρα και να πούμε ότι πρέπει να έχετε φτάσει σε αυτό το επίπεδο πριν περάσετε στο επόμενο και έτσι θα είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ενώ το benchmark χρησιμοποιείται στη διαδικασία προσχώρησης για να ανοίγουν και να κλείνουν διάφορα κεφάλαια, ε, συχνά προσθέτοντα και διμερεί ζητήματα. Ενώ ε, το benchmark υποδηλώνει κάτι περισσότερο από ε, ένα επίπεδο, είναι κάτι τελείω διαφορετικό, είναι περισσότερο ποιοτικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν ο σχόλιο γι' αυτό και για να περάσω και στην παρατήρηση για τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα που έκανε η κυρία Όμεν Ρόιτε και ξέρω ότι ασχολείται πολύ με τα θέματα των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας. Ε, τα θέματα αυτά είναι όλο και περισσότερο στην επικαιρότητα ακριβώ ε, διότι αντιμετωπίζονται προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο περισσότερε δυσκολίε υπάρχουν στα κράτη-μέλη, τόσο πιο αβέβαιοι είμαστε για την εφαρμογή τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τόσο πιο δύσκολο είναι να καθορίσουμε σαφή πρότυπα για τι χώρε οι οποίε προσδοκούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία θα μπορούσαμε να πούμε κάλλιστα ότι ναι, θα πρέπει να έχετε ελευθερία του τύπου, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη και να ορίζονται οι δικαστές από κάποια ανεξάρτητη επιτροπή. Ε, ή ο καθένας να έχει το δικαίωμα του λόγου στην ελεύθερη κοινωνία σας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίσουμε και τα εσωτερικά μας τα ζητήματα και όσον αφορά τη, ε, τα πρότυπα των κρατών μελών που ανέφερε η κυρία Κοπά στην έκθεσή τη, ε, που είναι σημαντικό θέμα και θα πρέπει να συζητηθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά το θέμα είναι να δούμε και τι θέλουμε να δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω τη εφαρμογή τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη Συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτή τη στιγμή μας απασχολεί όλους η ευρωπαϊκή κρίση και μόλις κατευνάσει αυτή η κρίση θεωρώ ότι αυτό είναι το δεύτερο, το επόμενο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και για την εξωτερική μας αξιοπιστία προς τις χώρες που θέλουν να εντοχθούν αλλά και προς όφελος των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, για την υποστήριξή σας και ιδιαίτερα για την υποστήριξη ε, της ε, συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και τη κοινωνία των πολιτών. Χαίρομαι που η κυρία Κοπά το σχολίασε. Εγώ για να εξοικονομήσω χρόνο δεν ανέφερα τι κάνουμε σε διάφορες χώρες. Ε, ίσως όμως θα ήταν καλή ιδέα να διοργανώσουμε κάποια κοινή εκδήλωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολιτικό επίπεδο και την ΕΟΚΕ ε, σε επίπεδο ε, κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών εταίρων. Ε, είναι ε, πολύ σημαντικό το ότι ε, βλέπουμε πως σε πολλές πόνταξη χώρες τα συνδικάτα είναι αδύναμα. Προφανώς όλα αυτά εξαρτώνται από την ιστορία και την παράδοση. Οπότε και μέσω της ΕΟΚΙ και μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων μας μπορούμε να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να βοηθήσουμε στην βελτίωση. Η διεύρυνση το 2004 και το 2007 ήταν, ε, έγινε πολύ καλά ε, και ήταν ε, μια ένεση βιταμίνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω τη συνέχιση της διαδικασίας με τις χώρες που χτυπούν την πόρτα μας και πληρούν τα κριτήρια. Νομίζω ότι η έκθεση είναι πολύ επίκαιρη, κυρία Κοπά. Ευχαριστώ. Thank you. We have set up uh, the... Η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 6η Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Η κυρία Κοπά μετά θα διαπραγματευτεί με όλους όσοι υποβάλλουν τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε, για την παρουσία σας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 today as well? Yeah, it's 12.30 today. All right. I'm it starts again in the afternoon. But in the afternoon... Ladies and gentlemen, lassen Sie uns zu Tagesordnungspunkt 6 kommen. Περνάμε στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Έχουμε μια σειρά εργαλείων μεταξύ αυτών τη θέσπιση κοινών κανόνων και λεπτομεριών εφαρμογής των μηχανισμών για την εξωτερική δράση της Ένωσης. Έχουμε ένα πακέτο για την βελτίωση της διαφάνειας και της λογικής συνέπειας των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτόν τον τρόπο, μέσω αυτού του πακέτου, θα ε, έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την συνέχεια και τη συνέπεια μεταξύ όλων των εργαλείων που διαθέτουμε. Οι εισηγητές ήδη συναντήθηκαν μεταξύ τους και συμφώνησαν επί ενός χρονοδιαγράμματος για την υιοθέτηση της στρατηγικής και των στοιχείων που αφορούν όλα τα όργανα, όλα τα εργαλεία, συγγνώμη. με κοινή έκθεση για τους ε, κοινού κανόνες. Οι τροπολογίες ε, αφορούν διάφορα θέματα. Γι' αυτό οι εισηγητέ αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια οριζόντια προσέγγιση. Στην τελευταία. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν από την Κομισιό να προτείνει μια διευρυμένη χρήση των κατεξιοδότηση πράξεων για την περίοδο 14-20. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και οι προτάσεις η ε, κατεξότηση ε, προτάσεων, ε, δεν ε, σέβονται το ρόλο του Κοινοβουλίου. Η, το Κοινοβούλιο όμως είναι συν για τον προγραμματισμό των εργαλείων που θα δοθούν στην Κομισιόν κατεξοδότηση. Το Κοινοβούλιο δεν θέλει να κάνει μικροδιαχείριση, Γι' αυτό το λόγο όμω θα πρέπει να ελέγξει την όλη διαδικασία και η διαδικασία να έχει μεθόδου προφύλαξη. και ε, αυτό θα γίνει μέσω των ε, κατεξοδότη πράξεων. Το στατικό πρόγραμμα και τα έγγραφα τα οποία καθορίζουν τι προτεραιότητε, του στόχου, τα αποτελέσματα και τη χρηματοδότηση σε γενικέ γραμμέ θα πρέπει να υιοθετούνται ω κατεξοδότηση πράξη. Το, ο τύπο των εγγράφων αυτών μπορεί βέβαια να προσαρμοστεί στο κάθε όργανο σε ό,τι αφορά τις ε, ε, της πράξης ε, ε, προβλέπεται ότι το ετήσιο πρόγραμμα θα ε, εφαρμόζεται, θα υλοποιείται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας ε, τα υπόλοιπα έγγραφα μέσω Συμβουλευτικής Επιτροπής. Δεύτερον, συνεργασία μεταξύ των εργαλείων. Η η προβλέπει ότι αν η αναδιαιτία έκθεση της Κομισιόν θα αξιολογεί την ε, συμπληρωματικότητα μεταξύ των οργάνων, μεταξύ των εργαλείων. Τρίτον, ανάγκη αξιολόγησης του αντικτύπου όλων των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αντίκτυπος αυτός θα πρέπει να αξιολογείται επαρκώς επί τη βάση σαφών δικτών που θα έχουν οριστεί για την αξιολόγηση κάθε εργαλείου. Τέταρτον, οι πολίτες της δικαιούχες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορούν να καταλάβουν το αποτέλεσμα των πράξεων, των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Είναι θέμα ορατότητας. Γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί ε, μια ε, στοχευμένη πολιτική ενημέρωση του κοινού ε, η οποία θα πρέπει μάλιστα να παρακολουθείτε σε ό,τι αφορά τα αποτέλεσματά τη. Πέμπτον, όπου είναι δυνατόν, οι θέσει των οργάνωσεων τη κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με διαφανή τρόπο για την εφαρμογή την υλοποίηση των προγραμμάτων. Έκτον, η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να δίδεται με βάση προτεραιότητες, σαφείς στόχους, κριτήρια απόδοσης, διαφάνεια και ε, κανότητα ε, λογιστικού ελέγχου. Έβδομον, αυτή η συμμετοχή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απαιτεί τα, μη, ε, τα όργανα που δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμοί μη ευρωπαϊκοί θεσμοί θα ε, ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μέχρι το τέλος, 2000, μέχρι το τέλος περίοδου 2014-2020 θα πρέπει ε, να γίνει προσαρμογή των χωρών οι οποίες λαμβάνουν την ενίσχυση στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα κοινή συζήτηση με τους άλλους ηγητές και συνεισηγητές. Νομίζω ότι ε, ε, αποτελεί προϊόν συνένεσης. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπέρμαν να πάρει το λόγο. Είναι ο εισηγητής για την ΔΕΒΕ. Είναι πολύ σημαντικό η ΔΕΒΑ να συνεργάζεται στενά με την ΑΦΕΤ. και για το κείμενο βέβαια, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Έτσι ενισχύουμε την ε, θέση και της ΔΕΒΑ και της ΑΦΕΤ. Ο κ. Μπέρμαν. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη κάνατε τις ρομαντικές σας ε, εξαγγελίες για την παθιασμένη συνεργασία ε, μεταξύ των δύο επιτροπών. Δεν θα τα επαναλάβω. Να μην γίνω και υπερβολικά ποιητικός, αν και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, εγώ είμαι συγγητής ε, για το DCI στην Επιτροπή ΔΕΒΑ. Η Επιτροπή μου επέτρεψε να με ορίσει και εισηγητή για την γνωμοδότηση για τον κανονισμό και το CIR και συμφώνησαν οι επιτροπέ ότι πρέπει να ε, λειτουργήσουμε συνδεδεμένε συνδεδεμένες επιτροπές. Ε, υπάρχουν αρκετέ ε, συνεδριάσεις, υπήρχαν αρκετέ συνεδριάσει ε, με το προσωπικό και για το CIR, αλλά και για να δούμε πώ ακριβώ οι διατάξει που συμπεριλαμβάνονται στο CIR θα επηρεάσουν τα μεμονωμένα ε, εργαλεία. Και ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικέ αυτέ οι συνεδριάσει. οδήγησαν σε ένα κοινό όρομα και κοινέ τροπολογίε. Η δική μου γνωμοδότηση έχει ολοκληρωθεί, θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή, στι 4 Ιουνίου. Η Επιτροπή ψηφοφορία, θα λάβει χώρα στι. 18 και 19 Ιουνίου. Ε, βεβαίως και κοίταξα την ε, έκθεση του κυρίου Μπρόξ. Η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Σχεδόν όλες οι τροπολογίες ε, που προτείνονται στην ΑΦΕΤ ε, υπάρχουν και στο δικό μου σχέδιο έκθεσης, πολλές φορές και με ταυτόσιμη διατύπωση. Σε γενικέ γραμμέ, οι πιο συγκεκριμένε θέσει μου και τροπολογίε έχουν σχέση με την εισαγωγή των εξή αλλαγών. Έξι σημεία αφορούν. Πρώτον, να καταστεί σαφέ ε, ότι υπάρχει διαχωρισμό μεταξύ των προγραμματικών αποφάσεων αφενό και των εφαρμοστικών αποφάσεων αφετέρου. Ο κύριος Μπρόκ το εξήγησε ήδη, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Είναι σαφέ όμω ότι ο Έμιλ Μπρόκ και εγώ έχουμε υποβάλει τροπολογίες για να εισαγάγουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Ε, και των όσων είπε στην διάσκεψη των Προέδρων ε, που εντόπισε τα στοιχεία που θα πρέπει να παρακολουθούμε τους στόχους, την επιλογή προτεραιοτήτων, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ε, ενδεικτική ε, κατανομή χρηματοδότηση για κάθε πρόγραμμα. Δεύτερον, ε, υπάρχει μια σειρά τροπολογιών μόνο για τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το DCI. Η επιλεξιμότητα ODA. Οι συνθήκες που ορίζουν ότι μια ενέργεια μπορεί να ε, θεωρηθεί... Ε, να ανήκει σε μια κατηγορία βοήθειας και στήριξης. Και μετά σε, σε κάποιες ε, ίσον τροπολογίε τροπολογίε, ενισχύω την ε, σημασία των, ε, των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, όπως είπε και ο, κ. στην εισαγωγή του. Χρειάζεται υποχρέωση από, από πλευράς Επιτροπής να υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσματα. Τέταρτον, κάποιε τροπολογίε τείνουν να περιορίσουν την διακριτική ευχαίρεια τη Επιτροπή. Η Επιτροπή προτείνει ε, μεγάλη διακριτική, περιθώριο διακριτική ευχέρεια, παρόλο που υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει ευελιξία ε, για την Επιτροπή για να ανταποκρίνεται ε, στην αλλαγή των καταστάσεων, των εξελίξεων σε αυτή την περίοδο. Όμω χρειάζεται και μια ισορροπία μεταξύ ευελιξία και κοινοβουλευτικού ελέγχου για την χρήση αυτών των κονδυλίων. Πέμπτον, το τελικό κομμάτι των τροπολογιών αφορούν τα άρθρα για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Ε, ε, ε, προκαλεί προβλήματα αυτή η διατύπωση στο κείμενο της Επιτροπής. Οι αναπτυσσόμενες χώρες που ανήκουν στο G20 δεν πρέπει, λέει, να έχουν πρόσβαση στους διαγωνισμούς που γίνονται υπό τον DCI υπό το εργαλείο εταιρικών σχέσεων. Εγώ ε, κοίταξα το... Το, το ε, υπάρχει διάκριση μεταξύ ε, μελών και μη μελών του G20 και έτσι αποκλείοντας κάποιε από τι αναπτυσσόμενε χώρε είναι κάτι απαράδεκτο. Γιατί ε, έρχεται σε αντίθεση με την ίδια την ε, πολιτική δέσμευση τη Ένωση. Το έκτο ε, σημείο. Ε, μεγαλύτερη μου, μεγαλύτερος μου είναι να διατηρήσω στις νομοθετικές προτάσεις τα ωφέλη που αποκομίσαμε πριν από έξι χρόνια. Όταν ε, διαπραγματευτήκαμε τα ε, υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα. Όπως ξέρετε, το τρέχον μέσω επιτεξιακής συνεργασίας είναι ένα από τα κύρια ε, μέσα που συζητούμε στο πλαίσιο των μεμονωμένων των επιμέρους μέσων. Υπάρχουν ήδη συμφωνίες που έχουν συναυθεί πριν από έξι χρόνια και από ό,τι φαίνεται η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις που αλλάζουν κάποιες από αυτές τις συμφωνίες. Αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι αποδεκτό. Θα σας δώσω τρία παράδειγμα. Πρώτον, ε, το κατόφλι που τίθεται. Ένα οικονομικό ε, κατόφλι ε, που έχει οριστεί και έχει και είναι ιδιαίτερα αυξημένο, πάει στα, στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πολύ ψηλό ποσό συνήθω για ένα μεμονωμένο project. Για να υπάρξει λοιπόν μια ελαφρύτερη εντό εισαγωγικών ε, διαδικασία. Έτσι αποκλείεται αυτό το πρόγραμμα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα έχουμε τα 10 εκατομμύρια ω κατόφλι και πρέπει να παραμείνει έτσι. Ε, η συμμετοχή ε, του κοινοβουλίου στου ελεγκτικού μηχανισμού πρέπει να παραμείνει σε... και δεν πρέπει να διαγραφεί από τον νέο κανονισμό. Και τώρα μια μικρότερη σημασία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να εξακολουθήσει να συνδέεται στην Διαχειριστική Επιτροπή. Πρέπει να συμμετέχουν όποτε συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, σε προγράμματα, σε project. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ο εισηγητή για το μέσο προενταξιακή βοήθειας εκ μέρους του κ. Πάσκου, ο οποίος είναι ο σκιώδη εισηγητή σας. Θα αναφερθώ στο μέσο προενταξιακής βοήθειας ε, το απόγευμα, πιο συγκεκριμένα. Ελπίζω η σκιά του κυρίου Πάσχου να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να σας καλύψει κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό το μέσο λοιπόν και τον κοινό κανονισμό εφαρμογή. Ο κύριο Πάσκου καταρχήν θα ήθελε να σα ευχαριστήσει για τη μεγαστή συνεργασία που είχατε με του κοιόδη εισηγητής των διαφόρων πολιτικών ομάδων και για το γεγονό ότι τα πιο σημαντικά ζητήματα για του σοσιαλιστέ και δημοκράτε ελήφθησαν υπόψη και τα έχετε συμπεριλάβει στις τροπολογίες που καταθέσατε και πιο συγκεκριμένα ε, μας ενδιαφέρει η εξέλιξη της κοινωνίας των πολιτών, το γεγονός ότι τα έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού είναι πράξεις εξουσιοδότηση επομένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης συμμετέχει εξίσου και το γεγονός ότι οι τοπικές και περιφερειακές ε, αρχές και ε, οι κοινωνικοί εταίροι λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ενθαρρύνονται προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία είναι κάτι το οποίο στόχο έχει να αυξήσει την προβολή της χρηματοοικονομικής στήριξης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και κάποιες μικρολεπτομέρειες και κάποιες αλλαγές που ίσως θα ήθελαν να κάνουν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Ε, μπορεί να καταθέσουν και σχετικές τροπολογίες. Το πρώτο αφορά τις τοπικές αρχές και το γεγονός ότι θα θέλαμε να συμμετέχουν περισσότερο ως δικαιούχοι της στήριξης ε, και θα μπορούσε να υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα ε, για την χρηματοοικονομική βοήθεια των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ώστε να είναι όχι μόνο αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τι επιχορηγήσει, αλλά είναι και αυτοί οι οποίοι υποφελούνται των έργων σε περίπτωση που απαιτείται. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα μέσα όπου μπορούμε να το ε, εφαρμόσουμε και συμβαδίζει και με το στόχο να συμμετέχουν περισσότερο οι κοινωνίε και όχι τόσο τα κράτη ω κράτη. Δεύτερον, ο κύριος Πάσκου και η πολιτική μας ομάδα θεωρεί ότι κάποιες από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για τον προπολογισμό, η τροπολογία 18 και η τροπολογία 20, υπερβαίνουν τα όσα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να μας οδηγήσουν σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία, πράγμα που μπορεί να δυσχεραίνει φυσικά και την χρηματοδότηση. Αυτό βεβαίως ε, χρήζει περαιτέρω συζήτηση θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε κάποιες διατάξεις που ε, διασφαλίζουν ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέσων όσον αφορά τους στόχους που προκύπτουν από τις συγκεκριμένε πολιτικές και τη στρατηγική Ευρώπη 2020, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του κλίματος. Τώρα, όσον αφορά τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, θα μπορούσαμε ίσω να ενισχύσουμε τη διατύπωση, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αρχή τη εταιρική σχέση σε όλη τη διαδικασία. Αυτό μπορεί να μα βοηθήσει να υποστηρίξουμε περαιτέρω τη δημοκρατία και τι συμμετοχικέ κοινωνίε, να δημιουργήσουμε καλύτερα στοιχεία επιτόπου και να ενθαρρύνουμε χώρε ε, να ξεκινήσουν διάλογο ώστε να περιλαμβάνονται όλοι. Εκ μέρου του κυρίου Πάσκου, όπω σα ανέφερα στην αρχή, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω, κύριε Μπροκ, για το γεγονό γεγονός ότι ε, λάβατε υπόψη όλους και τις ιδέες των σκιωδών εισηγητών και θα το πω και το απόγευμα, αλλά ως εισηγητές ε, για το μέσο προενταξιακής βοήθειας θα ήθελα να πω ότι ε, αυτή η ιδέα του να αντιμετωπίσουμε τα πάντα ως δέσμοι και να είμαστε πιο συντονισμένοι για όλους τους μηχανισμούς και κοινού εφαρμοστικούς κανόνες, κατά την άποψή μου μέχρι τούδε είναι υποφελής και ελπίζω ότι ε, και κατά τη διάρκεια της υποβολής και του συντονισμού ε, των τροπολογιών που μπορεί να προκύψουν από όλο τον εφαρμοστικό κανονισμό θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τη διαδικασία ώστε να μην υπάρχουν διαφιλονικούμενες αποφάσεις ε, για το κάθε μέσο στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία να σχολιάσω έναν δύο πραγματάκια παρόλο ότι έχουν γίνει ήδη αρκετά σχόλια. Ε, γίνεται λόγος για 30 εκατομμύρια. Μας φαίνεται αρκετά μεγάλο ποσό ε, το μηχανισμό σταθερότητας ε, μιλούσαμε για 20 εκατομμύρια τώρα προσθέθηκαν και άλλα 10 θα έλεγα ότι 20 είναι το ελάχιστο το μέγιστο το 30 μου φαίνεται υπερβολικό μια πρόταση σχετικά με την πρόληψη συγκρούσεων. Μια ανάλυση των συγκρούσεων θα μπορούσε να ενταχθεί σε όλα τα όργανα σε όλα τα εργαλεία που έχουμε και ενδεχομένως να συμπεριληφθεί και στην έγκαιρη, στον έγκαιρο προγραμματισμό. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη την πρόληψη των συγκρούσεων στον προγραμματισμό. Μετά για το άρθρο 6. που προβλέπει το δότηση προγραμμάτων εισαγωγών, κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν. Γι' αυτό λόγο θα ήθελα να διαγραφεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τους δείκτες αξιολόγησης, θα ήθελα να μου πείτε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα αυτό πρακτικά. Μετά για το άρθρο 17 ε, αναφέρεται μάλλον ε, αναφέρεται πότε θα ξεκινήσει ο κανονισμός αλλά όχι πότε θα λήξει. Ε, δεν θα πρέπει να συνδέεται με το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα, δηλαδή να λύγει το 2020. Το είπε και ο Σβέρμερ, νομίζω. Ευχαριστώ. Κύριος Κατσίν. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία, αλλά ιδιαίτερως για την προσπάθεια του να συντονίσει τα οριζόντια θέματα όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και για την ε, κοινή στάση επέναντι σε οριζόντια θέματα. Υποστηρίζουμε αυτή την κοινή προσπάθεια, την κοινή προσέγγιση και πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική μας θέση συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε επί στρατηγικών ε, γράφων προγραμματισμού ε, που θα υιοθετηθεί μέσω ε, κατεξοδότηση πράξεων. Τα υπόλοιπα έγγραφα θα μπορούσαν να υιοθετηθούν με την άλλη με κατεφαρμογή πράξης. Ε, ορισμένες πτυχές της EIDHR θα τις δούμε χωριστά, αλλά να αναφερθώ τρία θέμα, σε τρία θέματα που χρειάζονται περισσότερο προβληματισμό σε οριζόντιο επίπεδο. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την ορατότητα και την επικοινωνιακή πολιτική, ένας γενικός κανόνας μπορεί να είναι προβληματικός, διότι σε μερικές περιπτώσεις η δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την EIDHR ε, πρέπει να είναι ε, ε, κρυφή, ε, μυστική για να ε, μην θέσουν, σε κίνδυνο. Δεύτερον, το, η μέτρηση της, του αντικτύπου. Η IDHR λειτουργεί πολλές φορές σε δύσκολες συνθήκες, οπότε είναι δύσκολο να αξιολογηθεί πάντα το αντίκτυπος. Θα πρέπει να σκεφτούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τι σημαίνουν αυτοί οι δείκτες Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τον προπολογισμό, χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο να το εξετάσουμε και να δούμε αν σύμφωνουμε πλήρω. Το απόγευμα θα δούμε την κατάσταση με τον κ. σχέση με την IPA. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος το κοινοβούλιο να περιθωριοποιηθεί. Κάτι θα ήταν πραγματικά λάθος. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ορατότητά μας ιδιαίτερως σε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αρχικά θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για αυτή την ε, ολοκληρωμένη έκθεση. Είναι σαφές ότι τα, τα μέσα εξωτερικής ε, δράσης πρέπει να συνάδουν με τις ε, αξίες της Ένωσης και τις προϋποθέσεις που θέτει και το Κοινοβουλίο μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει και οι δικαιούχοι να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας η δυνατότητα πιθανών δικαιούχων να χειρίζονται τα κονδύλια με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να λυθεί υπόψη. Επιπλέον, φορείς της κοινωνίας των πολιτών στις ε, χώρες δικαιούχου πρέπει να ε, συμμετέχουν στη δικασία φαρμογής υλοποίηση αυτών των μέσων και κατά την ε, σύνταξη των κανόνων Αυτές οι οργανώσεις πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτά τα project που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριο Σαραζά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τα σχόλια που ακούσαμε από τους διάφορους εισηγητές Προφανώς το βασικό στοιχείο συζήτησης τις επόμενες εβδομάδες ε, θα είναι το θέμα των καταξουσιοδότησης πράξεων και τα ε, έγγραφα προγραμματισμού. Με τα χαράς βεβαίως να συζητήσουμε και θέματα προβολής και συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών φορέων ακόμα και εσωτερικώς οι συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο έχουν προχωρήσει από τότε που έγινε για πρώτη φορά η υποβολή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα ποια ήταν η θέση της Κομισιόν όμως. Ήταν τόσο σαφής και περιεκτική. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε όλο. Ίσως την επόμενη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει μια πιο μακροσκαλή, μια πιο σαφή και πιο επικοδομητική ε, απάντηση. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία άλλωστε. Πάντα ελπίζω, διότι εξ όσων κατανοώ εγώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τις υπόλοιπες επιτροπές, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να μην το καταλαβαίνει αυτό ποτέ και αυτό είναι ένα από τα βασικά μας προβλήματα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητούμε. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή που θα συνενώσουμε τις δυνάμεις μας με άλλους. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, δρά όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ παρόλα αυτά. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 14 Ιουνίου ε, στις 12 η ώρα. Συμφωνείτε όλοι. Ωραία λοιπόν. Κλείνει αυτό το ζήτημα. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Δημιουργία μέσου σταθερότητας να δώσω το λόγο στην κυρία Μπράντνερ, που είναι η συγγήτρια. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το μέσο σταθερότητα έχει συζητηθεί επανειλημμένω εδώ στην Επιτροπή μα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλαμβάνω τα είδη υποθέντα. Και απλώς θα ήθελα να υπενθυμίσω την, ε, κατά την άποψή μου, πολύ επιτυχημένη ακρόαση που κάναμε, η οποία μας ε, βοήθησε να δούμε τι κάνουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το μέσο σταθερότητα, πώ εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ένα-δυο πράγματα λοιπόν από πλευρά μου και κατόπιν ε, θα ακούσω ιδιαίτερα προσεκτικά του συναδέλφου που σίγουρα έχουν κάποια πράγματα να πούνε και κάποιοι από αυτούς ε, μου έχουν δώσει και την άποψή τους ε, τις τελευταίες εβδομάδες. Καταρχάς να σας πω ότι ε, συζητήσαμε απλώ τα οριζόντια ζητήματα ε, μόλις τώρα. Ε, κάποια είναι τροπολογίες στο μέσο σταθερότητα. επομένως δεν θα τα εξηγήσω τώρα αναλυτικά. Πολλά από αυτά αφορούν τις πράξεις εξουσιοδότηση. ούτε σε αυτά θα αναφερθώ. υπάρχουν συγκεκριμένε τροπολογίες από αυτό. Καταρχάς, και το είπα και στο παρελθόν, υπάρχει το θέμα του τίτλου. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η σταθερότητα αποτελεί δυσκολία για κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα την Τουρκία και το Μεξικό, που δεν θέλουν να θεωρούνται ασταθείς χώρες και υπήρχε πρόβλημα στη χρήση αυτού του μέσου για τις χώρες αυτές, ε, το ίδιο και για την ε, Αραβική Άνοιξη, όπου τελικώς ε, διαπιστώθηκε ότι επειδή εμείς είχαμε το δικό μας το μέσο σταθερότητας ε, και υπήρχε μία σύνδεση με την προηγούμενη πολιτική μας που θεωρούσαμε ότι η σταθερότητα βρίσκεται υπεράνω άλλων αρχών όπως είναι η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, δημιουργήθηκε κάποια ε, πρόβλημα να έχουμε ένα μέσο πρόληψης για παράδειγμα, πρόληψη που θα περιλαμβάνει τα πάντα. Ε, αν έχετε οποιαδήποτε πρόταση καλύτερη, είμαι διατεθειμένη να την ακούσω, δεν έχω κάποια αιμονή με το συγκεκριμένο τίτλο. Θα ήθελα απλώς ο τίτλος να αντικατοπτρίζει καλύτερα τι ακριβώς ε, σημαίνει αυτός ο μηχανισμός. Δεύτερο τώρα, για το πεδίο εφαρμογής. Προσπάθησα να προσπαθήσω να έχω τα αρκετή ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα να δίνω και κάποιες στρατηγικές κατευθύνσεις για το προς τα που θα θέλαμε να οδεύσει αυτό το ο μηχανισμός. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάσουμε την ευελιξία και ταυτόχρονα να έχουμε μια στρατηγική και να είμαστε επικεντρωμένοι κάπου σαφώς για την πολιτική μας. Προσπάθησα λοιπόν να περιορίσω λίγο το πεδίο εφαρμογής στα όσα δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο μέσο. Όπως είπαμε και προηγουμένως και αναφέρθηκε και στην ε, πρόταση, να συμπεριλάβουμε κάποιες δράσεις για τις ε, φυσικές καταστροφές και τις καταστροφές που προκαλεί ο άνθρωπος. Και φυσικά για τις ε, ε, φυσικές, φυσικές καταστροφές σε γέννη υπάρχει το ΕΚΟ για τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Αλλά ορισμένες ανθρωπιστικές κρίσεις μπορεί να κλιμακωθούν και να γίνουν κρίσεις ασφάλειας που διακυβεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια σε μια χώρα και στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτά δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε με το ΕΚΟ. Επομένως θα ήθελα να το περιορίσουμε και να αναφερόμαστε σε ασφαλ... Ε, απειλές για την ασφάλεια που προκύπτουν, που απορρέουν από τις φυσικές καταστροφές. Να μην θέλουμε δηλαδή να αποκλείσουμε και φυσικές καταστροφές, ε, να καλύπτονται αυτές από το μέσο σταθερότητας, αλλά να μην αναφερόμαστε αποκλειστικώ και μόνο σε ανθρωπιστικές κρίσεις, αλλά σε πιθανά δυνητικά προβλήματα ασφάλειας. Κατόπιν, για τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ε, μέτρα για την καταπολέμησή της, η Επίτροπος Βάλτνερ ε, κάποτε είχε υπογράψει μία δήλωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και από εκεί και πέρα στη συνέχεια ε, ότι εκπρόσωπος η κυρία Άστον, η, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, την επιβεβαίωση. Και αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικοί μηχανισμοί για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Υπάρχουν, για παράδειγμα, από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου πολύ καλέ κατευθυντήριε γραμμές Θα ήθελα λοιπόν να αναπτύξουμε και εμεί αντίστοιχε κατευθυντήριε γραμμέ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και το αναφέρω, το αναφέρω ε, ως παράδειγμα στο άρθρο μου, αλλά δεν θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να έχουμε αυτό το οποίο σας ανέφερα ως παράδειγμα. Θα ήθελα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη έχουν δικές τους κατευθυντήριες γραμμές, θα μπορούσαμε ίσως να εγκρίνουμε απλώς και τις δικές τους. Επόμενο σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2001 έχει ε, μία έννοια για τη διαμεσολάβηση και το διάλογο και ε, θεωρώ ότι είναι καλό το, η καλή έννοια αυτή και θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και εδώ. Δεν νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει δυσκολίες βέβαια. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία για τα μικρά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό. Ε, είναι πολύ σημαντικό ε, να πούμε ότι το μέσο σταθερότητας θα πρέπει να χρηματοδοτεί την καταστροφή αυτών των ε, όπλων το Συμβούλιο θεωρεί βέβαια ότι αυτό είναι εκτός πεδίου εφαρμογής ε, της κοινοτικής μεθόδου. Εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο χρήσιμο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ή τουλάχιστον είναι πολύ χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις μετά από σειράξεις να βρούμε πού βρίσκονται αυτά τα όπλα και να τα καταστρέψουμε. Ε, είναι βέβαια πολύ δαπανηρό αυτό. Ε, έχω προσθέσει ότι θεωρώ ότι εκεί μπορεί να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα ε, και να υπάρχει διαμάχη με το Συμβούλιο. Τώρα, για τα οριζόντια ζητήματα της οργανώσης της κοινωνίας των πολιτών, επί παραδείγματι, υπάρχει ένα σημείο μου στο οποίο θα ήθελα να ενισχυθεί αυτός ο ρόλος, ε, ιδίως για την αξιολόγηση μετά την υλοποίηση των μέτρων που χρηματοδοτεί το μέσο σταθερότησης. Όσον αφορά τώρα τον χρηματοοικονομικό φάκελο, εκεί υπάρχουν δύο σημεία που αφορούν τα χρήματα φυσικά. Και όπως είπα και προηγουμένως στη συζήτηση που μόλις κάναμε, θα ήθελα από τα 30 εκατομμύρια να ξαναπεράσουμε στα 20 εκατομμύρια, που ήταν το ποσό που είχαμε από τον προηγούμενο κανονισμό, Να μειώσουμε λοιπόν από τα 30 στα 20, δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες και μετά υπάρχουν τα κατεπήγοντα μέτρα. Εκεί θα ήθελα να αυξηθώ ή το ανώτατο όριο από τα 65 στα 70. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να κρατήσουμε και την ευρύτερη έννοια των φυσικών καταστροφών και αν όντω γίνει αυτό θα χρειαστούμε περισσότερα κονδύλια για να καλύψουμε και αυτό. Και θα ήθελα να διευκρινίσω ε, και για τα ποσοστά τι γίνεται για το άρθρο 4 και το άρθρο 5, το οποίο δεν τα, είχαμε όμως, ε, δεν τα έχουμε όμως αυτό στον κανονισμό, αλλά τα είχαμε στον προηγούμενο. Είχαμε κάποιες τροπολογίες από την Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, τις οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους τις έλαβα υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Gracias, presidente. Hemos trabajado muy estrechamente συνεργαστήκαμε στενά με την κυρία Μπράτνερ για να ρυθμίσουμε τα του κανονισμού περί σταθερότητας. Ε, συμφωνούμε με τα όσα προτείνει κατά βάση, εκτός από το τελευταίο σημείο. Τροπολογία 49. Τροποποίηση του άρθρου 13 της πρότασης κανονισμού. Σε ό,τι αφορά την αύξηση από το 65% στο 75% του ποσοστού για τις δράσεις του άρθρου 3 δεν θα μας δημιουργούσε πρόβλημα. Η Κομισιόν θα υπολογίσει πόσα χρήματα χρειάζεται για αυτό το κομμάτι των δράσεων. Όμως, η αύξηση για τις δράσεις υπό τα άρθρα 4 και 5, αύξηση δηλαδή από το 5% στο 15% είναι τόσο μεγάλη που θα πρέπει πρώτα να το δούμε με την Κομισιόν και με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, διότι αυτό θα σήμαινε τετραπλασιασμό των δράσεων. Και αν δεν είχαμε περιορισμούς, δημοσιονομικούς ε, περιορισμούς, δεν θα υπήρχε ζήτημα, αλλά υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί. Οι δράσεις υπό το άρθρο 4 αν αυξηθούν ε, θα πρέπει να μειωθούν οι δράσεις ε, που καλύπτουν από αλάθρα, για παράδειγμα το 5. Αυτό σημαίνει ότι θα έμενε χωρίς ε, προστασία του, μέτρου, του μέσου αυτού δράσεις όπως αυτή εναντίον της πειρατείας ή της ασφάλειας θάλασσα. Αν δεν έχουμε αρκετούς πόρους για τις δράσεις του άρθρου 5 ε, τέτοιου είδους ε, δράσεις, για παράδειγμα εναντίον της πειρατείας, ε, θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν μόνο από στρατιωτικά μέσα. Όμως, η δική μας άποψη είναι ότι με αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει να προσθέσουμε μια άλλη ε, ε, μια άλλη αντιμετώπιση του θέματος σταθερότητας, όχι μόνο στρατιωτική αντιμετώπιση. Συνεπώς θα ήθελα να το ξανασκεφτείτε, να ξανασκεφτείτε αυτήν την αύξηση από 5% στο 15% για τα μέτρα υπό το άρθρο 4. Ζητήστε αύξηση, αλλά ή μην πείτε σε τι ποσοστό ή αν πείτε ποσοστό μειώσετε, μειώστε το ποσοστό στο 7% αντί για 15% για παράδειγμα αλλά όχι τετραπλασιασμό του αφηρημένου αυτού στοιχείου του κανονισμού. Το μέσο αυτό είναι το πιο πολιτικό μέσο πραγματικά που έχει ως ε, στόχο την εξασφάλιση ενός αφηρημένου αλλά πολύ πολύτιμου αυτού της σταθερότητας. Οπότε είναι δύσκολο εκ των προτέρων να πούμε πού θα διοχετευτούν όλα τα ποσά και θα πρέπει να καλύψουμε όλο το φάσμα των δυνατών δράσεων. Ε, μην αυξήσουμε τόσο πολύ το ένα κομμάτι και αφήσουμε ακάλυπτο άλλο κομμάτι που ενδεχομένως θα αποδειχθεί ακόμα πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρέντερ Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μπρέντρινάρ για την συνεισφορά της. Το μέσο σταθερότητάς της έχει σαφέστερους στόχους σχέση με το παρελθόν. Στρέφεται περισσότερο προς ε, ένα μέσο που επικεντρώνεται στην ασφάλεια. Με, ε, διαγράφοντας τους ε, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους. Το πρόβλημα όμως εδώ είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης, της ευελιξίας και της δημιουργίας συνδέσεων ε, ανάμεσα στο μέσο για τη σταθερότητα και άλλων ε, μέσων ε, εξωτερικής ε, δράσης. Θεωρώ ότι η κοινωνική και η οικονομική πλευρά θα πρέπει να διατηρηθεί στο μέσο σταθερότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν μιλούμε για την επίλυση και αποτροπή, ε, η αποφυγή κρίσεων. Είναι ένας επιτυχής μηχανισμός ε, στην, όταν ε, πρόκειται για την ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε μια ακρόαση εδώ και οι πυρογνώμονες κατέστησαν σαφές ότι το μέσο σταθερότητας ήταν ε, ένα μέσο έκτακτης ανάγκης, σχεδιασμένο για διαφορετικές καταστάσεις και επομένως ήταν θεμελιώδης σημασία ε, η ευελιξία. Όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση από άλλους μηχανισμούς, ε, καλείται ο μηχανισμός σταθερότητα να ανταποκριθεί στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Από την άλλη, θεωρώ ότι το μέσο σταθερότητας θα μπορούσε να αποτελέσει δίωδο ε, προώθησης ε, των αναπτυξιακών πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί δικαιούχοι ε, χαιρετίζουν την ευελιξία ε, του μέσου και θα πρέπει να παραμείνει αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ. Βίλε Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που έκανε στην έκθεση. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα ήθελα να φέρω. Προς το παρόν θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε μια ε, συγκεκριμένη τροπολογία που προβληματίζει ιδιαίτερα ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αναφέρομαι στην τροπολογία 49 Ε, που σχετίζεται με το άρθρο 13. Θεωρούμε ότι αυτή η προτινόμενη τροπολογία θα δημιουργούσε πολύ μεγάλη ανισορροπία μεταξύ των ε, διαφόρων ε, πολιτικών του μέσου και τη κατανομής των κοντελίων για να διασφαλίσουν ε, την αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία του μέσου. Να σας υπενθυμίσω ότι η χρηματοοικονομική κατανομή για, για τέτοια μέτρα της ανάγκης ε, έχει τεθεί στα 73% ε, ενώ για άλλες μορφές είναι στο 5% ή στο 22% για την αποφυγή κρίσεων. Η προτεραιότητα τροπολογία θα αυξήσει ε, το, την κατανομή για το νέο άρθρο 4 από το 5% στο 15%. Στην πράξη αυτό αντικατοπτρίζει ε, σχεδόν 40%, 400% μάλλον ε, αύξηση αυτή η αστρονομική αύξηση θα ε, οδηγήσει σε δυσανάλογη χρηματοοικονομική κατανομή ε, για ορισμένα στοιχεία, δηλαδή για την πλευρά της αποφυγής κρίσεων, ε, που δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς. Εμείς θεωρούμε ένα τέτοιο τεράστιο ποσό δεν είναι σε καμία περίπτωση απαραίτητο για τους στόχους που προτείνονται. Παράλληλα και κατά συνέπεια αυτής της αύξηση, η τροπολογία θα μειώσει την κατανομή για το άρθρο 5 που όπως ξέρετε έχει ως στόχο την ε, επίλυση άλλων ε, ε, ζητημάτων το 22% στο 5%. Θα ήθελα να σε πιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι με μια τέτοια μείωση των κονδυλίων για τέτοιες παγκόσμιες προκλήσεις θα δημιουργηθούν προβλήματα και ανισορροπίες. Προβλέπεται επέκταση του άρθρου 5 σε νέου τομεί ε, παρέμβαση. Ο πραγματικό αντίκτυπο του άρθρου τη τροπολογία 49 είναι ότι θα έχουμε τρει-τέσσερι φορέ ε, μεγαλύτερα κονδύλια για κάποιου ε, τομεί από όσα χρειάζονται, ενώ για άλλου τομεί πολύ λιγότερα. Ε, σε επιχειρησιακού όρου αυτό σημαίνει ότι εμεί και εδώ, συμπεριλαμβάνω και την Επιτροπή, δεν θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πραγματικό ε, αντίκτυπο τις ε, ε, οικουμενικές απειλές όπως είναι ε, η, εμπορία ανθρώπων, η καταπολέμηση της πειρατείας και πολλοί άλλοι τομείς. Δεν θα επιτεύχουμε του στόχου λοιπόν σε αυτού του τομεί. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι σε θέση να επιτύχει του στόχου που έχει θέσει μαζί και με τι δράσει CFP, ECI, ENI για αυτού του λόγου καλούμε την ΑΦΕΤ και τα μέλη τη να επανεξετάσουν την συγκεκριμένη τροπολογία περιθμών 49. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Ντόιλ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Αρχικά θα ήθελα να στηρίξω απολύτω ε, τον ε, συνάδελφο από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης, ιδίω σε ό,τι αφορά την ε, κατανομή κονδυλίων για τα νέα άρθρα 4 και 5. Θεωρούμε ότι η αύξηση του ποσού για το άρθρο 4 στο 15% για τους, ε, για τις οργανώσεις οικοδόμησης δυναμικού είναι μια αύξηση ε, πέραν ε, του χρήσιμου. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω λόγω της ικανότητας απορρόφησης. Ε, στους ε, τομείς που καλύπτονται το άρθρο 5 έχει ήδη αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να υπάρξει απορρόφηση τέτοιων κονδυλίων και δεν πρέπει να το μειώσουμε. Αυτό θα γινόταν αν εγκριθεί αυτή η τροπολογία. Προτείνουμε λοιπόν να μείνει το κείμενο ως έχει την Επιτροπή. Να πούμε μόνο τουλάχιστον 65% για το άρθρο 3 για την ανταπόκριση κρίσεων για να διατηρηθεί μια ευελιξία για την ανταπόκριση στις ε, μελλοντικές εξελίξεις στα κονδύλια που θα κατανεμηθούν για τις δραστηριότητε από το άρθρο 4 και 5. Μερικές έχουμε παρατηρήσει. Στην τροπολογία 25 η Επιτροπή προτείνει μια δεύτερη επέκταση έξι μηνών, παράταση έξι μηνών. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όταν πρέπει να ε, ανασταλούν οι ενέργειες λόγω πολιτικών εξελίξεων και να υπάρχει δυνατότητα ε, επανεκκίνησης σε μεταγενέστερο στάδιο χωρίς επιπλέον ε, κόστος. Στην τροπολογία 28 Εκεί η Επιτροπή προτείνει τη δυνατότητα υιοθέτηση μέτρου χωρίς πρώτερη διαβούλευση σε εξαιρετικέ ε, περιπτώσει. Εάν ε, προσθέσουμε το με πρώτερη διαβούλευση, τότε ουσιαστικά έρουμε τον ε, χαρακτήρα της πρότασης. Το σενάριο που φαντάζομαι εγώ είναι, για παράδειγμα, ο που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε μια κρίση στη Συρία, για παράδειγμα, τότε υπάρχουν προσυμφωνημένες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από μια τέτοια ομάδα επαφής. Αν στο τέλος υπάρχουν συστάσεις ε, για παράδειγμα για, έναν, ε, για στήριξη ενός διεθνούς ε, δημοσιολαβητή, τότε είναι σημαντικό να μπορεί ο εκπρόσωπος να, να μιλήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να επιστρέψει και, και να διαβουλευθεί. Σε τέτοιες ε, περιπτώσεις θεωρούμε ότι υπάρχει μικρός κίνδυνος να υπάρξουν πραγματικές διαφωνίες από τα όσα θα έλεγε η Επιτροπή, είπατε εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος. Ε, ακούσαμε και κάποιες θέσεις στις 8 Μαΐου για την δυνατότητα ανταπόκρισης σε φυσικές καταστροφές ή και ανθρωπογενείς καταστροφές. Αυτό υπερβαίνει τα όσα μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε την σταθάνεια ή να αποφύγουμε τι αστάθειε. Δεν συνδέεται μόνο λοιπόν με συγκεκριμένε ε, ενέργειε, αλλά και για το, με το έργο τη ανοικοδόμηση. Και αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ε, ε, οικοδόμηση τη σταθερότητα. Να μην επιθέλετε σε λεπτομέρειε, αλλά 52, 53 και 58 και εκεί θα θέλαμε να επεξεργαστεί διατύπωση επειδή ακριβώ ε, ο κανονισμό για το μέσο σταθερότητα ε, προσδιορίζει ότι πρόκειται για ένα μέτρο ε, έκτακτη ανάγκη, όταν πραγματικά τίποτα άλλο δεν μπορεί να ε, δώσει χρηματοδότηση. Δεν θα αξιοποιήσουμε αυτό το μέσο για, για, για κάτι το οποίο μπορεί να καλυφθεί από άλλα μέσα. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριος... Ευχαριστώ Ζητώ συγγνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια αλλά με την έκθεσή μου στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, που είχε ταυτόχρονη συζήτηση με το θέμα αυτό, δεν μπορούσα να απουσιάσω από την Επιτροπή και ήρθα τώρα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είμαι θετικά διακείμενος στην ε, πρόταση της κυρίας ε, Μπραντνερ ε, και δέχομαι και αυτή την αλλαγή του τίτλου και θα ήθελα να προσθέσουμε και κάποια στοιχεία τα οποία ίσως θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες τροπολογίες στη συνέχεια. Ο σκιώδης εισηγητής ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Όπως είχα πει και στην πρώτη συζήτηση που κάναμε για το θέμα αυτό, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες πτυχές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξακολουθούν να φαίνονται ότι δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη την καινοτομία που αποτελεί η γέννηση αυτού του μέσου, αλλά και η ίδια συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία μας σωθεί προς την πιο συνεκτική χρήση των διαφόρων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν προσπαθεί να επιτύχει τους συνήθεις στόχους τους και να τηρήσει τις βασικές της αξίες και να υπάρχει μια ε, συνεκτική εξωτερική δράση. Ε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο ορισμός που έχουμε αυτή τη στιγμή στο άρθρο 1 σημείο 2α είναι παροχημένος κατά πάσα πιθανότητα, διότι συνδέει το μέσο σταθερότητας με τη δυνατότητα να επιτρέψουμε την ε, πολιτική της Ένωσης ε, Ανάπτυξης και ε, Συνεργασίας. Ναι, είναι ακανή και αναγκαία συνθήκη, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό δεν συνοψίζει τους ευρύτερους στόχους της Ευρώπης ε, και αυτό άλλωστε ε, ε, προτείνει και η ίδια η συγγήτρια όταν ζητά να αλλάξει ο τίτλος. Θα πρέπει λοιπόν να δεχτούμε πλήρως το νέο θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά τη δημιουργία αυτού του μέσου. Όσον αφορά τώρα το θέμα της κατανομής των πόρων. Συμφωνώ με την αύξηση του ορίου για το άρθρο 3, του ελαχίστου ορίου, διότι στην ουσία αυτό είναι ο συγκεκριμένο ρόλος του μέσου σταθερότητα. Νομίζω ότι η κυρία Μουνίθ Ντεορκίθα έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να διευκρινίσουμε την ελάχιστη κατανομή που έχουμε μεταξύ των άρθρων 3 και 4. Ίσως θα μπορούσαμε εδώ να συνδυάσουμε την πρόταση της εισηγήτριας με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία ίσονο σημασίας, αλλά ε, πέραν των όσων σας ανέφερα, σε γενικές γραμμές ε, είναι θετική η στάση μου για την πρόταση της κυρίας Μπραντνερ. Απομένει το θέμα της διαχείρισης των παραρτημάτων. Δηλαδή, ε, αυτή η νομική αλλαγή που περνάμε από τη συναπόφαση στις πράξεις κατεξουσιοδότηση ε, και εδώ ε, να συμφωνήσω με τα όσα από ό,τι έμαθα είπε ο κύριος Μπροκ ότι υπάρχει δηλαδή ανάγκη να επικαιροποιήσουμε τις πράξεις κατεξουσιοδότηση και να δράσουμε με βάση το πνεύμα της συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι θα ήταν το ίδιο αλλιώς αν να ξαναμένουμε στη διαδικασία της συναπόφαση, ακόμα και για τα πιο συγκεκριμένα σημεία που έχουμε στα παρατήματα 3, 4 και 5. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι έκθεση που θα μας ενώσει αντί να μας διχάσει. Είναι πολύ ε, θαρρυντική η δουλειά του εισηγητή. Το μέσο σταθερότητας είναι κρίσιμο προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθάει σε περιπτώσεις κρίσης. Χρειάζεται επίσης να συμμετέχει πιο καθαρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία, δηλαδή να ενημερώνεται, να ζητείται η γνώμη του και να, να λαμβάνονται υπόψη τα ψηφίσματά του και οι γνωμοδοτήσεις του. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί μια συνεπή συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν και την Περισσία Εξωτερική Δράση ο συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνει χώρα. Και η πράξη δείχνει ότι θα πρέπει να έχει και επίσημη βάση ε, προκειμένου να δώσει αποτελέσματα. Μερικά ερωτήματα. Στις τροπολογίες 55, 63 και 65 γίνεται αναφορά ή μάλλον διαγράφηκε η αναφορά στην δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε όμως ότι σε περιπτώσεις κρίσεων οι επιδημίες έχουν διασυνοριακές συνέπειες. Συνεπώς η δημόσια υγεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ε, σε ε, καταστάσεις που επικρατούν μετά τις συγκρούσεις. Ε, επίσης πολύ συχνά έχουμε την διασπόρα ε, εικονικών ε, ψευδοφαρμάκων. Επίσης γίνεται μία αναφορά, μάλλον διαγράφηκε η αναφορά στις, ε, ε στις θεομηνίες που πλήττουν παράκτιες περιοχές. Ε, θα ήθελα και αυτό να επιστρέψει το κείμενο. Κυρία Μπράντνερ. Θα απαντήσω στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Ε, η συνεργασία είναι πολύ χρήσιμη σε ό,τι αφορά την κατανομή την οποία αναφέρατε πολλοί από εσάς. Η αύξηση από 65% στο 70% είναι ε, ένα ποσό λιγότερο από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Παλιότερα είχαμε 73, συνεπώς λιγότερα από, τα, από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως είπε ο κ. το, η ομορφιά αυτού του μέσου ε, είναι η ευελιξία του. Οπότε η, μείωση, η θεώρησα ότι η μείωση από το 73 στο 65 ήταν πολύ και γι' αυτό λόγο επέστρεψα στο 70 διότι καλύπτουμε και θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, ανθρώπινης προέλευσης, καταστροφές κλπ. Ε, πώς είναι να το να προσθέτουμε δράσει και να μειώνουμε τον προπολογισμό. Ε, αυτά για το θέμα τώρα της προετοιμασίας και της πρόληψης κρίσεων. Το άρθρο λέει ότι θέλουμε να προλάβουμε τις κρίσεις και είναι ο καλύτερος τρόπος για την άποψή να ξοδεύσουμε τα χρήματά μας. Γιατί αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αν έχουμε ένα μόνο ευρώ, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτός είναι η πρόληψη και η προετοιμασία για τις κρίσεις. Ιδιαίτερα σε περιόδους λιτότητας, καλό είναι να προλαμβάνουμε αντί να ακολουθούμε τα γεγονότα. Και στο μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο περισσότερα χρήματα γίνεται για να προλαμβάνουμε και να προετοιμαζόμαστε για κρίση. Οπότε από στρατηγική πλευρά θα πρέπει να σκεφτούμε πού θέλουμε να ποντάρουμε τα χρήματά μα. Και όπω είπε η κυρία Μουνιό, αν είχαμε πακτολό χρημάτων δεν θα είχαμε πρόβλημα. Αλλά δεδομένου ότι έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμού, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια μας για πρόληψη και όχι για εκ των υστέρων δράση. Είναι λοιπόν μια στρατηγική στάση αυτή, να τη συζητήσουμε βέβαια. Νομίζω όμως ότι όλα τα ποσά που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη είναι πολύ λιγότερα από ό,τι θα χρησιμοποιούσαμε ε, αν δρούσαμε αργότερα για την ίδια περιοχή. Ας δούμε το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Ιεμένη κλπ από δημοσιονομική ε, πλευρά είναι νομίζω πολύ συνετό. Τώρα για τι μακροπρόθεσμες απειλέ. Ε, είναι πράγματι μια μείωση εδώ πέρα που κάπου πρέπει να γίνουν, να ε, πράγματι θα έπρεπε να, να, να αποφύγουμε αυτή τη μείωση, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο να αυξήσουμε το συνολικό ποσό για το μέσο για τη σταθερότητα ας προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το συνολικό ποσό του IFS. Και ο Σπρίντερ έφυγε, είπε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το μέσο αυτό και για αναπτυξιακή πολιτική. Όχι, ε, δεν θέλουμε ε, να ε, έχουμε επικαλύψεις. Η, χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, οι πόροι μας είναι λίγοι, οπότε θα πρέπει να τους ξοδέσουμε εκεί που δεν υπάρχουν άλλα μέσα για να εξασφαλίσουν τους στόχους μας. Σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση, Λέει το άρθρο ε, να υποστηριχθούν οι δράσεις για την έναρξη της ανοικοδόμησης και βασικών ε, υποδομών, στέγαση κλπ. Καθώς επίσης και άλλα μέτρα για την επανεκκίνηση οικονομικής δραστηριότητας, αύξηση της απασχόλησης και της, του καθορισμού των ελάχιστων ε, ε, συνθήκων για την κοινωνική ανάπτυξη. Αυτά είναι που προτείνονται. Όχι, εγώ διαφωνώ. Αυτό έχει σχέση με την αναπτυξιακή ενίσχυση ε, για το μέτρο για την αναπτυξιακή συνεργασία. Ε, εκεί, στο DCI, υπάρχει ευελιξία δεν θέλω τα χρήματα της, ε, του μέσου για την, για τη σταθερότητα να χρησιμοποιηθούν για την ε, κατασκευή ε, οικειών. Λυπάμαι πολύ, διαφωνώ. Είναι λίγα τα κονδύλια που διαθέτουμε. Άλλα σχόλια από την Κομισιόν για την δεύτερη παράταση. Ξέρω ότι ζητήσατε την παράταση για τη φορά. Γιατί, γιατί δεν έχει λειτουργήσει η αναπτυξιακή συνεργασία ε, και η ECR. Ε, δεν νομίζουμε όμως ότι χρειάζεται αυτή η παράταση. Τα επιτυχή προγράμματα θα πρέπει να τα αναλάβει, να τα λάβουν τα ε, μακροπρόθεσμα προγράμματα, όχι το δικό μας. Το σύστημα μας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε θα λειτουργήσει. Και τα μακροχρόνια μέσα θα πρέπει να λάβουν, την ευθύνη, την ευθύνη των προγραμμάτων τα οποία δεν θα συμπεριληφθούν στο μέσο για τη σταθερότητα. Γιατί πάλι θα καταλήξουμε να μην έχουμε αρκετά χρήματα για, την, ε, για, τις, ε, για τις επίγουσες καταστάσεις. Αυτά νομίζω ήταν τα βασικά, τα βασικά σχόλια, σας απάντησα, για τη δημόσια υγεία ε, και για τα ψευδή φάρμακα. Ε, καθώς επίσης και τις ε, ανθρωπογενείς καταστροφές και τις θεομηνίες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με όλα αυτά, ε, αλλά δεν πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να έχουμε ένα μέσο για τις θεομηνίες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ εστιασμένοι. Δεν είμαστε η ΕΚΟ, δεν είμαστε η υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας και υπάρχουν και στην EDF και στο DCI ε, χρήματα που οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα. Δεν συνεργάζονται βέβαια μεταξύ τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα δικά μας ποσά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπράντλερ. Και εγώ θα ήθελα να σας υποστηρίξω να συγκεντρώνουμε χρήματα για τους σωστούς σκοπούς και όχι απλώς να είμαστε καλοί με όλους. Ελπίζω να ε, μπορέσετε να το σκεφτείτε αυτό στη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, να δείτε τι γίνεται μετά την καταστροφή. Η, η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 14 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή...